Uh, good morning everybody. I wonder if I can... Uh, we are waiting for the commissioner who is... Καλημέρα σας. <clears throat> Μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, καθίστε παρακαλώ. Και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε γιατί όπως είδατε είναι ιδιαίτερα εργόδες το πρόγραμμα σήμερα. Δεν θέλω να χρονοτριβήσουμε λοιπόν. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί ομιλητέ οι οποίοι θα λάβουν το λόγο. Θέλω να σα ευχαριστήσω καταρχήν για την παρουσία σα εδώ και είναι μεγάλη χαρά για μένα να χαιρετήσω και τον Έντουαρτ Κούσισνικ, ο οποίο είναι ο εισηγητή τη Επιτροπή μα για την έκθεση πρωτοβουλία μα σε σχέση με το μέλλον τη ευρωπαϊκή τυποποίηση. Αυτή είναι και η αρχοκοκαλιά τη σημερινή ε, ακρόαση η έκθεση αυτή του κ. Κούσισνικ. Σας υπενθυμίζω ότι είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας, αλλά έχει χαιρετιστεί ευρέως ως μια ευκαιρία θα συζητήσουμε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη μελλοντική τυποποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά εν ώψη της σημαντικής νομοθετικής πρότασης που θα μας υποβάλει η Κομισιόν στο τέλος του χρόνου δεν είναι ένα θέμα η τυποποίηση που έχει εξεταστεί επαρκώς κατά την απόψή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία και με την παρουσία όλων αυτών των εξεχόντων εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται στα θέματα της τυποποίησης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλόδεκτη ευκαιρία να εξετάσουμε το θέμα αυτό και ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχίσει και στο μέλλον. Χαιρετίζω επίση την παρουσία και των μελών του Κοινοβουλίου εδώ. Οι σκιώδεις εισηγητές μας θα έχουν και αυτή την ευκαιρία να λάβουν το λόγο στη συνέχεια και αν συμφωνεί ο εισηγητής, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα θέλετε, θα θέλετε να κάνετε τώρα τις αρχικές σας παρατηρήσεις ή θέλετε να λάβετε το λόγο αργότερα. 20 λεπτά να περιμένουν πάρα πολύ, λέει ο εισηγητής. <clears throat> Τρία λεπτά. Τρία λεπτά μπορώ να περιμένω. Ώσπου να έρθει και ο, και ο Επίτροπος, ο κ. Σταγιάννη, και να ακούσει τον εισηγητή μας. Μέχρι τότε μπορώ να σας πω ότι η συνεδρίαση αυτή κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, κάθε λέξη μας τρέχει στο διαδίκτυο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι θα λάβουν το λόγο, θα πρέπει να ξέρετε ότι μόλις ανοίξετε το μικρόφωνο σας θα εστιάσει απάνω σας μια διαδικτυακού χαρακτήρα κάμερα. Και πρέπει να χρησιμοποιείτε λοιπόν το μικρόφωνο που είναι στο δεξί σας χέρι για να λειτουργήσει σωστά και η κάμερα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι να έρθει ο Επίτροπος, εκτός αν έχουμε κάποιο άλλο θέμα να διεκπαιρεώσουμε. Uh, well, ladies and gentlemen, uh, Mr. Is, uh, just on his... Κυρίες και κύριοι, καταφτάνει ο κύριος Σταγιάννη. Οπότε να κάνουμε κάποιες ανακτήρες παρατηρήσεις και μετά θα περάσουμε στις πρώτες δηλώσεις των συναδέλφων. Παρακαλώ καθίστε. I know there were a number of breakfasts over the last two days around... Ξέρω ότι κάποιοι καθυστέρησαν στον πρωινό, στο πρωινό. Χαίρομαι πολύ που υπήρξε τόσο ενδιαφέρον και επίσης να πω ότι υπήρξε η... στο συνάντηση του πρωινού η συνάντηση ακριβώς η συζήτηση της ενδιάμεσης ομάδας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν ε, έχετε καθυστερήσει από το πρωινό αυτό θα βρείτε τα ανάλογα έγγραφα μπροστά σας. Να σας ενημερώσω τώρα για το πώς εξελίσσεται αυτή η έκθεση. Για το τελευταίο τρίμηνο του φετινού έτους και το επόμενο εξάμηνο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς για το πρόγραμμα της Επιτροπής. Είναι μεγάλη μας χαρά που επιτέλους έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο για την Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα. Καλώς ήρθατε κύριε Ταγιάννη. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι ότι η κυρία Κέπχαρτ ήδη εργάζεται για μια, πιστεύω, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση. Και αφού ακούσουμε και εσά σε αυτή την ακρόαση, θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση αυτή τον Ιούλιο, στην τελευταία μα συνεδρίαση πριν την θρηνή διακοπή. Στι 13 του μήνα δηλαδή. Μετά θα δούμε το σχέδιο της έκθεσης ε, στη συνάντησή μας του Σεπτεμβρίου και με τα μέλη και σκοπεύουμε στις 30 Σεπτεμβρίου να ψηφίσουμε σε επίπεδο επιτροπής και έπειτα τελική ψηφοφορία τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουμε και βεβαίω ελπίζουμε ότι έτσι θα συμβάλλουμε και στο έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Για να ξεκινήσει λοιπόν η συνεδρίαση. Καλωσορίζουμε και πάλι τον Επίτροπο που είναι αρμόδιο για αυτή την σοβαρότατη νομοθετική πρόταση στον τομέα τη τυποποίηση. Απλώ θα ξεκινήσω δίνοντα το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Κότσουσνικ και να, δώσω, και να συγχαρώ και τον κύριο Beauty ο οποίο ετοιμάζει μια σημαντικότητα γνωμοδότηση για μα εκ μέρου τη Επιτροπή Βιομηχανία, που θα επηρεάσει και αυτόν τον τομέα που συζητάμε τώρα από πολλές διαφορετικές σκοπιές, ιδίως τον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και των ε, νέων τεχνολογιών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή και μετά θα ακούσουμε βεβαίως ε, και την ομιλία του Επιτρόπου. Επίτροπε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε χρόνο και για ερωτήσεις από τους βουλευτές, αλλά θα εξαρτηθεί αυτό και από τους δικού σας περιορισμούς. Ευχαριστώ Μάλκον. Θα μιλήσω στα τσεχικά, <clears throat> που είναι η μητρική μου γλώσσα. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, <clears throat> ίσως ο Μάλκομ και εγώ είμαστε οι μόνοι που έχουμε την ευκαιρία να λάβουμε δύο φορέ το λόγο σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχουμε μια μεγάλη πίεση χρόνου και αυτό γιατί ήμασταν φιλόδοξοι, προσπαθήσαμε να προσκαλέσουμε όλου του εμπλεκόμενου στα θέματα τυποποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ακούσουμε τι απόψει του σε σχέση με την τωρινή κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μελλοντικέ προοπτικές τυποποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ξεκινήσω λοιπόν με ορισμένες ε, παρατηρήσεις. Είχαμε ένα πρόγευμα εργασίας πριν από δύο-τρεις μέρες και συζητήσαμε για τις επιτυχίες της διαδικασίας τυποποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι η τυποποίηση είναι ένα εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Είναι ένα μέσο το οποίο θα μας δώσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη προφανώς είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πολίτες μας. Και είναι ένα σημαντικό εργαλείο σε ό,τι αφορά την παροχή δημοσίων υπηρεσιών. Μπορεί να είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα έχουμε καλύτερο έλεγχο των δημοσίων υπηρεσιών και είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε μια αρρύθμιση από τη βάση και όχι εκ των άνω. Εγώ σκέφτομαι με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε την τυποποίηση πιο εναργή, πιο σαφή. Και έχω ένα παράδειγμα που σχετίζεται και με την Ιταλία. Πέραν των πολιτικών μου δραστηριοτήτων, εγώ και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες, προωθώ ένα νέο σπορ που λέγεται beach tennis. Δεν είναι beach volleyball. Μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Ένα νέο σπορ Αλλά παρά το γεγονό ότι είναι νέο σπορ, στην Βόρεια Ιταλία είναι περίπου 300.000 άτομα που παίζουν το beach tennis. Ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια και τώρα έχει διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι καθώς αναπτυσσόταν αυτό το σπορ υπήρχαν Ιταλικοί κανόνες, Αμερικάνικοι κανόνες, Αγγλικοί κανόνες και <clears throat> τα τελευταία τρία χρόνια οι κανόνες του beach tennis σε όλο τον κόσμο εναρμονίστηκαν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και για την Ευρώπη και για τους Ευρωπαίους παίκτες. Έχουν λοιπόν εναρμονιστεί κανόνες, επομένως όλοι παίζουν στα ίδια γήπεδα με τις ίδιες προδιαγραφές και με τους ίδιους κανόνες beach tennis. Υπάρχουν κανόνες για τις ειδικές ρακέτες που χρησιμοποιούνται στο άθλημα αυτό και αυτό φυσικά έχει ανοίξει νέες αγορές. Γιατί οι περισσότερες από αυτές τις ρακέτες παράγονται στην Ευρώπη, ιδίως στην ιταλια ή πέντε εταιρείε τις παράγουν, τις κατασκευάζουν. Με την ενοποίηση λοιπόν των κανόνων, οι ευρωπαϊκές ρακέτες εξάγονται στη Βραζιλία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, μέχρι και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Χάρη στην τυποποίηση λοιπόν αυτού του νέου αθλήματος, έχει προκύψει και μία πηγή καταναλωτών. Υπάρχει τώρα μια παγκόσμια ομοσπονδία παικτών του beach tennis η οποία πρότεινε και νέα νέα μπαλάκια τα οποία θα βοηθήσουν να παίζετε καλύτερα αυτό το σπορ. Σας λέω λοιπόν ότι έχει νόημα αυτή η τυποποίηση, αυτού του είδους η τυποποίηση ξεκινά από τη βάση και είναι ένας με τον οποίο μπορούμε να προωθούμε τα συμφέροντα της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος λοιπόν για την έκθεσή μας, όπως τονίστηκε και από τον Malcolm Harbour, είναι να εξεύρουμε μια ισορροπία μεταξύ της δραστηριότητας τυποποίησης από την πλευρά της Κομισιόν των εθνικών γραφείων τυποποίησης των καταναλωτών και των συμφερόντων τους και γενικά των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό είναι ο στόχος της δικής μου έκθεσης με τη συνεργασία των σχεδόν εισηγητών και είμαι έτοιμος να ακούσω τα σχόλιά σας για την κατάσταση και το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο Ρένχαρτ Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε κάποιες από τις ε, σκέψεις που έχουμε στην ε, Επιτροπή μας. Χαίρομαι επίσης που άκουσα και τον εισηγητή. Ε, είχα ένα πρωινό σήμερα όπου ο κύριος Γκουτσογιάννης από την Ευρωπαϊκό Γραφείο μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων ε, και χειροτεχνίας μας είπε πόσο σημαντική είναι η τυποποίηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είπε πως είναι ακόμη πιο σημαντική και από την έρευνα. Ένα από τα σημεία στα οποία δίνω έμφαση στη δουλειά μου μέχρι στιγμή είναι το πώς θα επηρεαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην τυποποίηση. Κατά βάση νομίζω πως όταν μιλάμε για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουμε τρεις λέξεις κατά νου. Κόστος, πολυπλοκότητα και συμμετοχή. Προφανώς υπάρχει κάποια εμπειρία στους εθνικούς οργανισμούς ε, τυποποίησης για να προσφέρουν πακέτα τυποποίησης ε, με μειωμένο κόστος. Νομίζω πως είναι πολύ καλή αυτή η προσέγγιση. Επίσης υπάρχει ανάγκη να παρουσιαστούν να παρουσιάζονται στο διαδίκτυο αποσπάσματα της ε, τυποποίησης έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να έχουν καλή πρόσβαση στις ε, προδιαγραφές που ίσως τις αφορούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και προφανώς μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά για να μειώσουμε την πολυπλοκότητα των προδιαγραφών πρέπει να φροντίσουμε στις αρχές του ΠΟΕ η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η σημασία και η αμεροληψία να, συμπε... να συμπεριληφθούν πλήρως ε, στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Και όσον αφορά την συμμετοχή υπάρχει μια συζήτηση είναι μια συζήτηση που αξίζει προσοχή. Υπάρχει εθνική συμμετοχή που θα μπορούσε να ενισχυθεί και από ε, συμμετοχή στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάποια από αυτά τα πράγματα συζητάμε στην Επιτροπή μου. Και τέλος, ένα πράγμα ακόμα. Θεωρούμε πως θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην υπόσχευση που θα μπορούσε να είναι το να μοιραστούμε τις ε, προδιαγραφές με διεθνείς εταίρους για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σε διεθνείς αγορές. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, που αναφέρατε κάποιους τομείς κλειδιά και θα επιστρέψουμε σε αυτούς. Ε, βεβαίως, ε, όπως ξέρετε, πρέπει τώρα να δώσουμε τον λόγο στον Αντώνιο Ταγιάννη, τον Επίτροπο βιομηχανία και επιχειρηματικότητα και χαιρόμαστε τώρα που έχει και τον τίτλο της επιχειρηματικότητα, αν και είναι δύσκολο να το προφέρει κανείς ακόμη στα αγγλικά. Αντώνιο πρέπει να σου το λόγο γιατί πρέπει να πας στη Νέα Υόρκη. Αλλά χαίρομαι που είσαι εδώ σήμερα το πρωί σε αυτή την ακρόαση εκπροσωπώντας την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε θα πρέπει να βιαστώ γιατί θα πρέπει να πάω και στο αεροδρόμιο για την πτήση μου προς Νέα Υόρκη, αλλά σήμερα έχουμε συνάντηση με τον κύριο Μπαν Κιμούν. Και τώρα θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Για το θέμα της τυποποίησης θέλω να ευχαριστήσω κατά πρώτον την δική σας επιτροπή, την Επιτροπή ΙΜΚΟ, που αποφάσισε να διοργανώσει αυτήν την ακρόαση, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται τις νέες αποφάσεις για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Για μέ λοιπόν, για το συνεργάτες μου και για τη γενική μου διεύθυνση, το να ακούσω αυτή τη συζήτηση είναι εξαιρετικής σημασίας. Εδώ εργαζόμαστε για την αναθεώρηση του συστήματος τυποποίησης και σκοπεύουμε να Υποβάλλουμε προτάσεις έως το τέλος του χρόνου. Η όλη συζήτηση καθώς και η έκθεση πρωτοβουλίας που επεξεργάζεται το Κοινοβούλιο θα είναι συνεισφορές καθοριστικές και για το δικό μας το έργο. Πριν συζητήσουμε το μέλλον, θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν, κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό των όσων έχουν γίνει ως τώρα. Το ευρωπαϊκό σύστημα είχε αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και φάνηκε ότι είναι ένα καθοριστικό εργαλείο για να ευνοήσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Υπό το φως αυτών των δεδομένων μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν επιτυχημένο το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης ως τώρα. Για να αναφέρω ορισμένους τομείς μόνον. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Εκεί απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Σε διεθνέ επίπεδο υπάρχει αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα ω προ τον ορισμό των προδιαγραφών και δεν πρέπει να μελούμε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα πολύ συχνά αφορά τομεί και περιοχέ παρέμβαση που δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί αρκετά. Και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση, έχουμε ξεκινήσει ένα σχέδιο αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματο τυποποίηση με δύο γύρους δημοσίων διαβουλεύσεων. Ασχοληθήκαμε με τα ΤΙΚ και επίσης ενδιαφερθήκαμε για όλα τα άλλα θέματα οριζόντιου χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα εξετάζουμε τα πορίσματα της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που ανέλαβαν το να παρουσιάσουν τη μελλοντική εξέλιξη του Ευρωπαϊκού συστήματο τυποποίηση με ορίζοντα το 2020. Και επίση φροντίζουμε να εντοπίσουμε τι αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα του μελλοντικού συστήματο και εδώ μιλώ για τι διαδικασίε τυποποίηση για τη χρηματοδότηση τη τυποποίηση σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτή η διαδικασία αξιολόγηση είναι καθοριστική σημασία για το πόσο θα μπορέσουμε να παρέμβουμε με τρόπο στοχευμένο και αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται, ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι πρέπει να υποφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα του ισχύοντος συστήματος. Αυτό το σύστημα παρουσιάζει πολλά σημεία ισχύω, τα οποία μας δίνουν ε, τα κατάλληλα θεμέλια για να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε περαιτέρω το όλο σύστημα. Ε, είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει βέβαια περιθώριο για βελτίωση για την εξωτερική διάσταση πρώτα απ' όλα. Στο διεθνέ επίπεδο θα πρέπει να προωθήσουμε την αριστεία του δικού μα προτύπου τυποποίηση σε διεθνέ επίπεδο. Όπω ξέρουμε, η Ευρώπη έχει ε, ένα σύνηθε ε, στρατηγικό πλεονέκτημα που καταφέρει να επιβάλλει παρά να υποστεί την υπεροχή των ε, προτύπων της. Έτσι θα καθοριστούν και οι ισορροπίε στι διάφορε αγορέ. Έτσι λοιπόν πρέπει να ισχυθεί ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των οργανισμών προτύπων και σε επίπεδο των διεθνών οργανισμών προτύπων, όπω του Διεθνού Οργανισμού για την Τυποποίηση. Θα πρέπει να σκεφτούμε και τους εμπορικούς φραγμούς, διότι μπορεί να παρουσιαστούν προσκόμματα στο εμπόριο λόγω της πρόβλεψης ε, εθνικών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε νομική υποχρέωση για όλους όσοι ετοιμάζουν πρότυπα και σε επίπεδο ΠΟΕ και στο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού, όπως είπε και ο συνάδελφος Μπουτικόφερ στην παρέμβασή του τώρα για την εξωτερική εσωτερική διάσταση. Και εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη η λειτουργία του συστήματός μας. Οι ευρωπαϊκοί φορέ τυποποίηση θα πρέπει να επιχειρήσουν να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες ώστε να δημιουργηθούν ε, δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τους. Επειδή οι πόροι που διαθέτουμε είναι περιορισμένοι σε αυτή την περίοδο της κρίσης, οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να επεξεργαστούν και να τελειοποιήσουν μέσα ανάλυσης και εξέτασης, τα οποία θα πρέπει να ε, ολοκληρώνονται και να έχουν περατωθεί πριν από την ε, διεξαγωγή ενός συγκεκριμένου προγράμματος τυποποίησης. Έτσι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις πρωτοβουλίες που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στον χώρο του εμπορίου και της αγοράς. Θα πρέπει να ανανεωθεί εδώ και να αναθερμανθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διεθνών οργανισμών τυποποίησης. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, θα πρέπει τα πρότυπα και διαδικασίε ανάπτυξη των προτύπων να είναι πάντοτε πιο προσβάσιμοι, ιδίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό είναι κάτι που σχολίασα και ο κύριος Μπούτικοφ. Αυτό θα είναι σπονδυλική στήλη τη ε, ε, για να αρθούν και τα προσκόμματα και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην πορεία της τυποποίησης. Θα πρέπει όλοι οι κανόνες ε, των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ε, εμπίπτουν στον τομέα της τυποποίησης. Επίσης, στον τομέα της καινοτομίας θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η τυποποίηση από την αρχή των διαδικασιών καινοτομίας προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη και η διάδοση της ίδιας της καινοτομίας Και αυτό και στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματο καινοτομία που θα παρουσιάσουμε μαζί με την Επίτροπο Γιώργαν Κουίν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για το νέο πρόγραμμα τυποποίησης. Για τα ΤΕΚ, όπως θύμισα στην αρχή της παρέμβασής μου, θα πρέπει να αποβεθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης παρακολουθεί και τις ε, συνεχείς εξελίξεις των προτύπων. Εδώ, στο δεύτερο μέρος των ΤΕΚ, θα πρέπει να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφο σε διεθνέ επίπεδο. Εάν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να δώσει ζωή στι νέε τεχνολογίε, θα πρέπει να μεγιστοποιήσει την ανταγωνιστικότητά τη στου διάφορου βιομηχανικού τομεί. Και θα πρέπει να είναι διορατική και να θέτει μακροπρόθεσμου στόχου σε αυτό το τομέα. για να αναλάβουμε και ρόλο επικεφαλής εδώ, πρωταγωνιστικό όπως επιθυμούμε. Θα πρέπει να ενσωματώνουμε όποτε χρειάζεται τα έγγραφα και τα πρότυπα που ετοιμάζονται από τα διεθνή φόρα και κονσόρσια και επίσης να εγκαθιδρύσουμε διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό της διατουργικότητας. Οι υπηρεσίες ε, λειτουργίας θα πρέπει να μπορούν να συνδυάζονται ώστε να ανταποκρινόμαστε στους κοινούς μας στόχους. Σε ό,τι αφορά το θέμα που για μένα είναι ιδιαίτερα προσφυλές της προσβασιμότητας ε, για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Θα πρέπει εδώ να συζητήσουμε τρία ζητήματα. Στο πλαίσιο του νέου πακέτου θα πρέπει να προβλέψουμε προδιαγραφές για την τυποποίηση που αφορούν ευαίσθητου τομείς. Ένα παράδειγμα, η πρόσβαση, η πρόσβαση για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες η προστασία των καταναλωτών για να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο κάλυψης του πολίτη. Εδώ θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία ε, εξεργασίας των, ε, των προτύπων ανάλογα και την ετοιμασία νέων προϊόντων. Επίσης τα περιβαλλοντικά πρότυπα είναι απαραίτητα λόγω χάρη για τη μέτρηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η τυποποίηση θα είναι μια αποφασιστική συμβολή και για τις πολιτικές που σχεδιάζουμε για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Περίπου 10% των Ευρωπαίων πολιτών υποφέρουν από κάποια μορφή αναπηρίας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι η διαδικασία γέρανσης του πληθυσμού αφορούν ε, το μέλλον της Ευρώπης, γιατί οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν. Επιπλέον, αξιολογούμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε δραστηριότητες τυποποίησης στον τομέα των υπηρεσιών. Στην πρόσφατη, στις πρόσφατες διαβουλεύσεις που είχαμε, ε, το σύνολο των ενδιαφερομένων έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ε, συμπερίληψη, συμπερίληψη των υπηρεσιών ε, κατεξοχήν των υπηρεσιών των μεταπολιτικών. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω την θέση του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με το θέμα αυτό. Για να ολοκληρώσω, να πω ότι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτά τα προβλήματα, ετοιμάζουμε ένα πακέτο ε, τυποποίησης, το standardization package. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, σκοπεύουμε να εγκρίνουμε το πακέτο αυτό τον μήνα Νοέμβριο. Το πακέτο αυτό θα αποτελείται από μια ανακοίνωση που θα καθορίζει το μελλοντικό όραμα της πολιτικής τυποποίησης με ορίζοντα το 2020 και θα εξετάζει τα βασικότερα θέματα τα οποία έθιξα και εγώ στη διάρκεια της ομιλίας μου. Οι αλλαγές αυτές στο νομοθετικό επίπεδο κατά πάσα πιθανότητα θα προβλέπονται από ένα ενιαίο έγγραφο, ένα κανονισμό. Ο κανονισμός αυτός θα υποκαταστήσει όλες τις νομοθετικές πράξεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο ό,τι αφορά την τυποποίηση και επιπλέον θα εγγυηθεί την καλύτερη υλοποίηση των πολιτικών τυποποίησης. Αυτή η λύση θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλλει στο να δώσω και μεγαλύτερη προβολή στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως βλέπετε είναι πολλά αυτά που έχουμε να κάνουμε και το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένει μια περίοδο συναρπαστική και γεμάτη προκλήσεις στο χώρο που σήμερα συζητούμε. Θα ήθελα λοιπόν να δείξετε ανοιχτό πνεύμα στη στα διάφορα θέματα που πρόκειται να συζητήσουμε, διότι όλοι οι συνεργάτε μου, τη γενική διεύθυνση και του δικού μου γραφείου, είναι στη διάθεσή σα. Επίση, θα αφήσω στον πρόεδρο Χάμπο το κείμενο τη παρέμβασής μου και τι προτάσει που έκανα ώστε να συμπεριληφθούν στα πρακτικά τη ακρόαση και βεβαίω θα είμαι στη διάθεσή σα. Δυστυχώ σήμερα δεν γίνεται γιατί θα χάσω την πτήση μου για τη Νέα Υόρκη. Εάν όμω θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε στην Επιτροπή πριν το καλοκαίρι, δηλαδή πριν την ε, υποβολή τη ανακοίνωση του όλου κειμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσουμε με του εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου για ένα τόσο σημαντικό θέμα, την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού μα τομέα και όπω υπογράμμισα και στην ομιλία μου, να δώσουμε συγκεκριμένε αποκρίσει σε όλου του Ευρωπαίους πολίτε. και κατεξοχήν στι ομάδε που είναι πλέον ευάλωτε και περιμένουν από εμά συγκεκριμένε απαντήσει. Οι τεχνολογικέ εξελίξει δεν θέλουμε να του αφήσουν ε, εκτός των, ε, της νέας πραγματικότητας. Αυτά από την πλευρά της Επιτροπής. Ε, με συγχωρείτε που δεν μπορώ να συμμετάσχω περαιτέρω στη συζήτηση, αλλά οι συνεργάτες με τη Γενική Διεύθυνση είναι στη διάθεσή σας για να σας ακούσουν και να αξιοποιήσουν και τις προτάσεις και τις συνεισφορές σας για τη μελέτη των δική μας των νομοθετικών μας κειμένων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Ήταν χαρά μας και πολύ σημαντικό που ακούσαμε το πώς ενδιαφέρεται προσωπικά ο για αυτό το σημαντικό τομέα και όπως τον ακούσατε να λέει ελπίζει το πακέτο της τυποποίησης να υιοθετηθεί το Νοέμβριο. Και, όπως είπα και πιο πριν, πριν έρθει, σκοπεύουμε να ψηφιστεί η έκθεσή μας τον Οκτώβριο αλλά βέβαια θα έχουν γίνει τα περισσότερα μέχρι τότε. Οπότε νομίζω πως έχουμε εδώ ένα καλό παράδειγμα στρατηγικής σκέψης της Επιτροπής μας, καθώς ε, θέλει βεβαίω να δημιουργήσει το πλαίσιο. Επίσης η κυρία Βάισενχόν ε, από την Κομισιόν είναι εδώ παρούσα και έχει λάβει σε αρκετές ε, συναντήσεις και θα είναι εδώ σήμερα αυτή και η ομάδα της και καλωσορίζω επίσης ε, Χόντα μέλη του Συμβουλίου ή των κυβερνήσεων των κρατών μελών που ξέρω πως επίσης δραστηριοποιούνται στο να υποβάλουν προτάσεις σε αυτόν τον τομέα. Οπότε περνάμε τώρα στους ε, προσκεκλημένους μας στο πακέτο που έχετε μπροστά σας. Κυρίε και κύριοι και κύριοι βουλευτές έχετε βιογραφικά όλων επειδή έχουμε λοιπόν λίγο χρόνο και πολύ ενδιαφέρον για αυτή την ακρόαση, έπρεπε να στριμώξουμε λίγο τους ομιλητές, αλλά ξέρω ότι θα σεβαστούν τον χρόνο και για να τους βοηθήσουμε θα δείχνει και ένα ρολόι η οθόνη. Οπότε, πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή τυποποίηση σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και έχουμε εκπροσώπους οργανώσεων που είναι στην καρδιά αυτής της διαδικασία. Και καλωσορίζω πρώτα απ' όλα τον Κέβιν ε, Μακίνλεϊ που είναι ε, αναπληρωτής γενικός γραμματέας στον ε, ΆΙΖΟ στη Γενέβη και Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας πως είχαμε μια πολύ επιτυχή αποστολή στην Γενέβη εξ ονόματο της Επιτροπής μας και επισκεφθήκαμε και τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και τον ΟΗΕ εκεί όπου θα πάει ο κύριο Σταγιάννη βεβαίως επισκεφθήκαμε τον ε, Οργανισμό Πνευματική Ιδιοκτησίας και τον ΠΟΕ οπότε θέλω να τον ευχαριστήσω δημοσίως ε, για το πώ μα καλωσόρισε όρισε και θα σας ε, παρακαλέσω να λάβετε πρώτον τον λόγο εξ ονόματος των προσκεκλημένων μας. Έχει τον λόγο. Μεγάλη χαρά που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και μπορώ να παρουσιάσω τις απόψεις της ISO και της IEC. Τι είναι καταρχήν αυτή η φορήση. Είμαστε διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη διεθνών προτύπων. Η IC είναι στον ηλεκτρικό τομέα και ηλεκτρονικό τομέα και η ISO ασχολείται με σχεδόν όλα τα άλλα θέματα κάτω από τον ήλιο, αυτοκίνητα, βίδες, κοινωνική ευθύνη, τα πάντα. Τόνισα ότι η ISO και η IEC είναι μη κυβερνητικοί φορείς και επίσης υπάρχει και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, η ITU, η οποία συνεργάζεται μαζί μας με στόχο να αναπτύξουμε παγκόσμια πρότυπα, τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις και τη σύγκληση των τεχνολογιών. Η ISO και η IEC έχουν την ίδια άποψη ότι πρέπει να υπάρχει μια συλλογική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία των μερών από 163 χώρες. Μέσω αυτών η Ευρώπη είναι πράγματι πολύ παρούσα που παίζει σημαντικό ρόλο και στους δύο αυτούς φορείς. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν μεγάλη διασύνδεση και με τα προγράμματα εργασιών της ISO και της IEC και με τον τρόπο αυτό με τις ρυθμίσεις αυτές υπάρχει μια στενή σύνδεση και με τη ΣΕΝ και ΣΕΝΕΛΕΚ. <clears throat> Ποια είναι λοιπόν τα ε, ζητήματα που συνδέουν την ε, ISO και την IEC με την τυποποίηση και τον υπόλοιπο κόσμο. Όλα αυτά γίνονται μέσω της συμφωνίας της Δρέσδης και της Βιέννης, για τις Δρέσδης για τη ΣΕΝ και ΣΕΝΕΛΕΚ και της Βιέννης για την ΑΕΣΥ και ΆΙΣΟ, που προβλέπουν την ε, υιοθέτηση των προτύπων αυτών από την Ευρώπη και επίσης και μηχανισμούς με τους οποίους άλλοι οργανισμοί μπορούν να εισαγάγουν ευρωπαϊκά πρότυπα, είτε με κοινέ δράσεις είτε με διεθνείς συμφωνίες. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό ανάπτυξης προτύπων ώστε να εξασφαλιστεί και η σύνδεση της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο. Κυρίως με τον τρόπο αυτό η ευρωπαϊκή προσέγγιση έχει επηρεάσει ιδιαίτερα θετικά την διεθνή δημιουργία προτύπων. Από τη δική μας οπτική γωνία της ISO και της IEC αυτές οι συμφωνίες είναι ιδιαίτερα καρποφόρες. Αλλά αυτές οι συμφωνίες επίσης βασίζονται στην ε, τωρινή βάση συμμετοχή στην IEC και ISO, δηλαδή επί τη βάση εθνικών ομάδων συμμετοχής. Εάν αλλάξει αυτή η βάση θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την, ε, τον τρόπο λειτουργία μας και ιδίως τη συνεργασία μας με τι ΣΕΚ και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις οι οποίε μπορούν να προκύψουν. Εδώ βλέπουμε τη σημασία των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίηση και των εμπλεκομένων στην ISO. Υπάρχουν οι ομάδε εργασίας που εκεί υπάρχουν περίπου 1.064 ηγέτες οι οποίοι διορίζονται από μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι περίπου το 53% όλων των τέτοιων ηγετικών θέσεων. Επίσης, οι προεδρίες επιτροπών είναι περίπου 52% και οι γραμματείες και αυτές 365 θέσεις, τα μισά, οι μισές προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική παρουσία, αν συγκρίνουμε και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΑΕΠ παγκοσμίω. <clears throat> Επίσης, η αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. Έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο στο χρόνο ανάπτυξης, 30% μείωση από το 2003 στην περίπτωση της ανάπτυξης προτύπων στην ISO και επίσης υπάρχουν άλλε βελτιώσεις οι οποίες θα προκύψουν ιδίω στι διαδικασίες της ISO. Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τεχνολογία. Έχουμε ένα σύστημα με πλατφόρμες στο διαδίκτυο, έχουμε διασκέψεις φωνητικού χαρακτήρα από απόσταση για τις συνεδριάσεις επιτροπών μεταξύ εμπειρογνωμόνων εταιρικέ σχέσεις με άλλους φορείς προτύπων και τυποποίηση είναι πολύ σημαντικά όταν γίνεται ένα έργο με πρόορη προετοιμασία, με πρώιμη μάλλον προετοιμασία και αυτό μας δίνει μια μεγαλύτερη ε, αποτελεσματικότητα και επίσης προωθούμε νέα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τις ε, εθνικές αντιπροσωπείες προτύπων και τους εμπλεκομένους. Τα διεθνή πρότυπα γίνονται ένα υπόδειγμα καινοτομίας. Οι πολιτικές μας και οι διαδικασίες ε, επιτρέπουν και προωθούν την καινοτομία μέσω των κοινών προτύπων και επίσης δίνουν την κατάλληλη πληροφόρηση προς καταναλωτές για καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αγορά. Επίσης τα νέα τεχνολογικά θέματα όπως η ανατεχνολογία, τα βιοκαύσιμα, κλιματική αλλαγή, βιοτεχνολογία, θέματα αηφορία είναι ζητήματα όπου η Ευρώπη έχει μια ιδιαίτερα μεγάλη παρουσία και ένα σημαντικό ρόλο. Υπάρχει ανάγκη να μπορέσουμε να έχουμε μια παρουσία στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης προτύπων, την παρουσία και των ακαδημαϊκών κύκλων. Η ISO, η IEC και η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών κάνουν μια τέτοια ακαδημαϊκή βδομάδα τον Ιούλιο στην Γενέβη και επίσης ο στόχος μας είναι να δείξουμε ποια είναι τα ωφέλη που θα προκύψουν για τη βιομηχανία από μια πιο διάφανη σύνδεση μεταξύ των ομάδων τυποποίησης ακολουθώντας την στάνταρ μέθοδο Roland Berger για που προβλέπεται στο σύστημα ISO. Επίσης μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια πρόσβαση στα πρότυπα αυτά. Εμείς δεχόμαστε τις βασικές αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού <clears throat> Εμπορίου για τα διεθνή πρότυπα. Επίσης θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των εμπλεκομένων και των εθνικών αντιπροσωπιών. Επίσης όλο και περισσότερο προχωρούμε σε μια φάση όπου είναι πάρα πολύ κέρια η συμμετοχή των εμπλεκομένων και αυτό φαίνεται και από τη Γενική μας Συνέλευση, η επόμενη θα είναι στον Σεπτέμβριο. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για αναθεώρηση από τη βάση και φυσικά τα πρότυπα αυτά πολλούνται και γίνεται η κεντρική τους διάθεση και από τον φορέα μας και από τα κράτη-μέλη. Είναι όλο και πιο διαθέσιμα τα πρότυπα αυτά και αυτό πρέπει να αυξηθεί έτσι περισσότερο. <clears throat> τα συστήματά μας βασίζονται λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία πώλησης γιατί είναι ουδέτερα και αποτελεσματικά μέσα ανάπτυξης νέων προϊόντων και φυσικά προωθούνται και από τις οργανώσεις των κρατών μελών. Το να υπάρχει απόλυτα ε, δωρεάν διάθεσή τους βέβαια είναι μια ιδέα, αλλά αυτό θα θέσει ίσως ένα αμφιβόλο την διατήρηση των φορέων μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ε, ευκαιρία αυτή να θέσω τα θέματα αυτά υπόψη σας και να σας πληροφορήσω για τις προοπτικές τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. thank you very much indeed, Kevin. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κέβιν, και είναι χαρά μας να σε καλωσορίζουμε εδώ. Είπες ε, κάποια σημαντικά πράγματα για το μέλλον και τις δεσμεύσεις ε, των κρατών ε, της κοινότητας και είμαι σίγουρος ότι θα αναφέρθουν αυτά μετά σε ερωτήσω. Ε, η επόμενη τώρα ομιλήτρια νομίζω δεν χρειάζεται παρουσίαση. Είναι η Έλενα Σαντιάγκο. Περνάει πολύ καιρό τελευταία στο Κοινοβούλιο και χαιρόμαστε γι' αυτό γιατί είναι πάντα βεβαίως έχει πάρα πολλά να μας πει και πάρα πολλές ε, πληροφορίες ε, στον ρόλο της ως ε, Γενικός Γραμματέας του ΣΕΝ και ΣΕΝΕΛΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή σας που μας δίνει αυτή την ευκαιρία γιατί πράγματι αυξάνεται έτσι ε, το πόσο φαίνεται η ευρωπαϊκή τυποποίηση που αποτελεί βεβαίω το μισό θα έλεγα πρόγραμμα εκπαίδευσης που κάνουμε. Είμαστε ένας πολύ δυναμικός οργανισμός. Θα ήθελα βεβαίω να είμαι όρθια αλλά δυστυχώς πρέπει να καθίσω εδώ πέρα δεν μπορώ να δω τις αντιδράσεις σας όταν μιλάω αλλά ως εργαζόμενη μητέρα με τρία παιδιά από 18 μήνες μέχρι 12 έτη ηλικία νομίζω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω και τα προβλήματα του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Τυποποίησης. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τις συστάσεις και θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω όλους ε, όσους παρακολουθείτε και εδώ μέσα και από το διαδίκτυο να μοιραστείτε αυτές τις συστάσεις και να τις υιοθετήσετε για να εκμεταλλευτείτε πλήρως το σύστημά μας. Απευθύνομαι πρώτα απ' όλα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργανά και τις αρχές ε, των κρατών μελών και σε όλους όσους ε, υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή τυποποίηση ή θεωρούν ότι μπορεί πράγματι να έχει μια προσθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία και να συνεχίσουν να στηρίζουν και να προωθούν το σύστημα ως έχει με την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ειδικού ε, που γνωρίζουν το θέμα και αυτοί συμμετέχουν στην κατάρτιση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και συμμετέχουν βεβαίως έτσι και είναι υπέρ του παγκοσμίου εμπορίου. Ακούσαμε και τον Κέβιν και υπάρχουν και εθνικές αντιπροσωπείες ε, που στηρίζουν την συμμετοχή όλων των ενδιαφέρομενων. Πώς μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία με το να επεκτείνουμε το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης σε νέους τομεί όταν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από αυτούς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τις προδιαγραφές. Και μπορούμε βεβαίω ε, να το προωθήσουμε περαιτέρω όταν, ε, είμα, έχουμε συνοχή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λέξη συνοχή. Η δεύτερη σύστασή μου είναι να υπάρξουν επίσημοι δεσμοί με την καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση. Και εδώ πέρα αναφέρομαι στα εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης ε, και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουμε σε οποιονδήποτε οργανισμό που βασίζεται στην γνώση στην Ευρώπη και μπορούμε έτσι να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματά μας πολύ πιο γρήγορα. Και βεβαίω όπως φαντάζεστε δεν θα μπορούσα παρά να συμπεριλάβω τα χρήματα, δίδυ χρημάτων και των δεν. Είναι σημαντικό αυτό για τις δραστηριότητες τυποποίησης. Χρειαζόμαστε λοιπόν οικονομική βιωσιμότητα. Θεωρούμε πως ε, σταθεροί κανόνες και χρήσιμοι προς τον χρήστη είναι κάτι το κρίσιμο για να προωθήσουμε τις αξίες του συστήματός μας. Θα προσπαθήσω τώρα να ορίσω αυτές ε, τις αξίες και μετά να σας δώσω κάποιους λόγους για το πώς ε, υποστηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. βεβαίω. σκοπεύουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ, αυτό είναι ήδη κτημένο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα τυποποίηση και τα εθνικά συστήματα αυτά, αλλά εμείς πάμε παραπέρα. Το σύστημα μα είναι ανεξάρτητο γιατί προσπαθούμε να μην έχουμε κάποιον με δεσπόζουσα θέση στις τεχνικές επιτροπές. Είναι καινοτόμο γιατί προσαρμοζόμαστε στις ε, κοινωνικές ε, και οικονομικές ανάγκες, έχουμε συνοχή, προσπαθούμε να μην έχουμε αλληλεπικάλυψη στις να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτά τα οποία παράγουμε. Δεν θέλουμε οι εταιρείε στην Ευρώπη που συμμετέχουν σε πολλές, ε, να συμμετέχουν σε πολλές τεχνικές επιτροπές για να έχουν τυχόν αντικρώμενα αποτελέσματα για να γιατί έτσι θα χάσουμε βέβαια την ανταγωνιστικότητα που είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημά μας. Πώς υποστηρίζουμε λοιπόν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Διαμορφώνουμε την ενιαία αγορά. Υπάρχει μία προδιαγραφή ίδια για 31 χώρες. Μιλάμε για πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Και υπάρχει μία προδιαγραφή Όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν οφείλουν να αποσύρουν τυχόν άλλες προδιαγραφές που είναι διαφορετικές. Αυτό βασίζεται στην γνώση γιατί οι προδιαγραφές παράγονται από τους ειδικού που ξέρουν το θέμα το οποίο τυποποιούν, γνωρίζουν τι συνέπειες θα έχει αυτό και πώς αυτή η προδιαγραφή θα μπορεί να εφαρμοστεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι κερδίζουμε από τη διεθνή διάσταση, έχουμε άμεση εμπλοκή στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης και χάρη στην τυποποίηση η Ευρώπη τοποθετείται στην παγκόσμια αγορά. Επηρεάζουμε και παίζουμε ηγετικό ρόλο στους τομείς στους οποίους μπορούμε γιατί έχουμε ε, την ε, ηγεσία στην τεχνολογία. Διασπείρουμε επίσης την πληροφορία και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί η καινοτομία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γνωρίζουμε πως πρέπει να βελτιώσουμε τη σχέση με την έρευνα και την ε, καινοτομία. Είναι λοιπόν κάτι το σαφές ότι μιλάμε, όταν μιλάμε για πρωτακαφές, μιλάμε για μεταφορά γνώσης. Μειώνεται το κόστος λοιπόν θέσης ενός προϊόντος στην αγορά και έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε και μια διαφοροποίηση για τις ευρωπαϊκές αγορές γιατί τα βασικά πράγματα καλύπτονται από την τυποποίηση, οπότε οι εταιρείε μας μπορούν να ασχοληθούν με τις καινοτομίε υψηλής αξίας για να μπορέσουν να κερδίσουν ποσοστό στην αγορά και βεβαίω διασφαλίζουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους ε, ανταγωνιζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε ανταγωνίζονται με ίσους όρους οποιαδήποτε άλλη μεγάλη εταιρεία όταν έχουμε τυποποιημένα προϊόντα ήθελα να επανέλθω τώρα στα ωφέλη για την ε, κοινωνία, γιατί υπάρχει εδώ πέρα και, υπάρχουν και τα κοινωνικά συμφέροντα τα οποία ενσωματώνονται. Αυτό γίνεται μέσω των εθνικών επιτροπών και φορέων τυποποίηση. Όποιο θέλει λοιπόν να έχει τη δυνατότητα να το κάνει, γιατί αυτό μπορεί να γίνει στην γλώσσα του. Εάν κάτι είναι το ε, αποτελεσματικό, ο κανονισμός ακολουθεί την τελευταία λέξη τεχνολογία και βρίσκουμε τρόπο να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία. Έχουμε επίση οικονομικό όφελο, έχουμε αποδείξει πω υπάρχει μια συνεισφορά 25% στην αύξηση του ΑΕΠ και βεβαίω επωφελούνται και οι καταναλωτέ και η κοινωνία γιατί όλοι ε, επωφελείστε από ασφαλή προϊόντα, φιλικά προ το περιβάλλον, που είναι προσβάσιμα και ανταγωνιστικά σε μια λογική τιμή για τον Ευρωπαίο καταναλωτή και αυτό γίνεται χάρη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ευχαριστώ πάρα πολύ. Well, thank you. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ δυναμική και σαφής παρουσίαση και μέσα στα χρονικά όρια, τα τυποποιημένα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο θέμα όπου έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και την καινοτομία και μιλάω περισσότερο για τις τηλεπικοινωνίες και την, ε, τις ε, τεχνολογίες πληροφόρησης. Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω τον Τζον Φίλιπς, τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της ε, Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Προτύπων Τηλεπικοινωνιών. Έπρεπε να φοράω και εγώ την γραβάτα μου του Ινστιτούτου. Αυτή φορά δεν είχαμε γραβάτα για τη ΣΕΝΕΛΕΚ, αλλά ελπίζω να μου δώσετε κάποια στιγμή. Τζον, χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που είσαι παρόν και μπορείς να αναφερθείς στο έργο της Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι η Σέγκη Ελέκ θα σας δώσουν επιτέλους αυτή τη γραβάτα που περιμένετε. Όταν μιλάμε για την τυποποίηση των ε, προτύπων τεχνολογιών και πληροφόρηση στην Ευρώπη είναι δύο θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχη βιομηχανίας σήμερα, <clears throat> πώς έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμή πρότυπα και πώς συνεχίζει να το πράττει. Δεύτερον, θα πρέπει να κατανοήσουμε ποιε είναι οι διαγραφόμενε τάσει. Μόνο τότε μπορούμε να δούμε ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά μια τυποποίηση φιλική προ το χρήστη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εξέλιξη που απαιτείται από το τωρινό σύστημα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε υποστήριξη αυτών των επιθυμητών χαρακτηριστικών. Αυτή θα είναι λοιπόν και η παρουσίασή μου σήμερα. Περνάω στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν, την τυποποιημένη διαφάνεια, η οποία αναφέρεται στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, οι οποίες υποστηρίζουν παγκόσμιες αγοράς. Η αγορά προωθείται από τους εμπλεκόμενους, που είναι πολλές φορές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επιχείρηση και το υποδειγματικό το υπόδειγμα επιχειρήν αλλάζουν με τρόπους που δεν προβλέπονται πάντα από τα πρότυπα και τα πρότυπα βέβαια δεν πρέπει να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η εξέλιξη. Οι παραγωγοί προτύπων θα πρέπει να υποστηρίξουν τη βιομηχανία τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και να βοηθήσουν στη δημιουργία οικονομικής αξίας. Αν αναδυφίσουμε την τα αποτελέσματα προτυποποίησης που ήταν σημαντικά στο παρελθόν, όπως είναι το ίντερνετ, το σύστημα ψηφιακών τηλεφώνων, τα νέα συστήματα για σταθερή τηλεφωνία, συστήματα τα οποία εξάλλου είναι σε κατάσταση σύγκληση σήμερα, το τεχνικό τμήμα της προτυποποίησης γίνεται σε σόρου σε, σε χώρους όπου δεν υπάρχει επίσημη πάντα συμμετοχή, είναι πιο άτυπη αυτή η διαδικασία και τα σώματα τυποποίησης που χρησιμοποιεί η βιομηχανία αυτή έχουν επιχειρηματικά μοντέλα που αντανακλούν τις προτιμήσεις της βιομηχανίας για να υπάρξει μια φτηνή παροχή προτύπων για να επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη του βιομηχανικού αυτού τομέα και να υπάρχει μεγαλύτερη επιρροή σε παγκόσμιο χώρο. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών πληροφορίας και πληροφοριών δεν μπορούν να αγνοηθούν είναι το γενικό πλαίσιο με στο οποίο πρέπει να λάβει η χώρα <clears throat> η διαδικασία προτυποποίησης. Η έτσι λοιπόν το Ινστιτούτο μας δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Χρησιμοποιεί τις ε, ε υπηρεσίες επιχειρηματιών, διοικητικών, ακαδημαϊκών για να επιτύχει το ρόλο της. Είναι ένα πάρα πολύ Επιτυχέ μοντέλο που χρησιμοποιεί και την παρουσία από μικρομεσαίες επιχειρήσει μέχρι μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και από κρατικούς φορείς, 25% των μελών μας έρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό οδήγησε σε μεγάλη επιτυχία, χάρη, το σχέδιο εταιρική σχέση για την τρίτη γενιά, το 3GBP, όπου υπήρξε μεγάλη συμμετοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. 70% των συμμετεχόντων ήταν από την έτσι και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη συστημάτων κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς και για δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα. Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι διαγραφόμενες τάσεις. Υπάρχουν τρεις κύριοι τομεί. Πρώτα, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας είναι πια πανταχού παρόντες στην καθημερινή ζωή. Υποστηρίζουν την κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και είναι και ένας μηχανισμός για άειλα αγαθά και άειλες υπηρεσίες. Δεύτερον, αυτό απαιτεί μία ε, διαφάνεια των τεχνολογιών αυτών για τους καταναλωτές και χρήστες που περιμένουν διαλειτουργικότητα, απόλυτη διαλειτουργικότητα πέρα των τεχνολογικών επιλογών. Τέλος, αυτή η πανταχού παρουσία των τεχνολογιών αυτών πρέπει να υποστηρίσει και πλήρη συστήματα για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που θα διαθέτουν αυτή τη διαλειτουργικότητα και γι' αυτό ζητά ακόμα περισσότερο από την προτυποποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα επίπεδα διαλειτουργικότητας τα οποία έχουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και έρχομαι τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Το σύστημα αυτό χρειάζεται να μετεξελιχθεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες τυποποίησης που ανέφερα και τις ανάγκες της βιομηχανίας. Να προσκαλέσει περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πλαίσιο αυτό και επίσης μεγάλες εταιρείες για να συνεργαστούν με αποτελεσματικό τρόπο. Αν κατανοήσουμε λοιπόν την ανάγκη να υπάρχει μια πλήρης διαλειτουργικότητα και πλήρης συστήματα παράδοσης υπηρεσιών και αγαθών, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε πια να περιμένουμε με λογικό τρόπο να υπάρχει μόνο ένας φορέας προτύπων ο οποίος θα καλύψει όλα τα απαραίτητα πρότυπα. Γι' αυτό χρειάζεται και συνεργασία μεταξύ φορέων προτύπων και το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης έτσι θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό ως εταίρος στα θέματα παγκόσμιας τυποποίησης. Μέσα στην Ευρώπη αυτές οι αλλαγές αποτελούν την πρόκληση που μας κάνουν να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρμόσουμε το σύστημα στην ανάγκη της βιομηχανίας. Πρέπει φυσικά να παραμείνουμε μέσα στο πλαίσιο των προτύπων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε και ένα ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίηση, το οποίο εξακολουθεί να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική μέσω ενό κατάλληλου συστήματο διακυβέρνηση τη καινοτομία και των προτύπων πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Η Ευρώπη να γίνει ένας αποτελεσματικός και φιλικός χώρος για τυποποίηση στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργήσει μια ευρεία βάση πλατφόρμα συνεργασίας για την τυποποίηση για τις τεχνολογίες αυτές και ιδίω να δώσει την δυνατότητα να υπάρχει πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοράς. Εγώ πιστεύω ότι η επιτυχία στην τυποποίηση είναι το να μπορέσει να δημιουργηθεί από τα πρότυπα αυτά μια κοινότητα συμφερόντων από τους εμπλεκόμενους στο βιομηχανικό τομέα και με τον τρόπο αυτό μπορεί ένα πρότυπο να ευδοκιμήσει. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η χρονική αλληλουχία των γεγονότων, να είναι έγκαιρη η δημιουργία αυτών των πρότυπων. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζει τι συνεργατικέ ενέργειε, όπω τα προγράμματα εταιρική σχέση που προαναφέρθηκαν και επίση θα πρέπει να συλλέξουμε την τυποποίησή μας και τα στάνταρ μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταλαμβαδεύονται στις βιομηχανίες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσης και το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει και η συμμετοχή ατύπων φορέων όταν αυτοί ακολουθούν τις προδιαγραφές μας. Θα πρέπει να επιτρέψουμε λοιπόν να χρησιμοποιηθούν τα πορίσματα αυτών των φορέων διαβούλευσης και στις δημόσιες προμήθειες και στη δημόσια πολιτική. Σίγουρα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς ε, συνεργασίας που επιτρέπουν την άμεση συμμετοχή των εμπλεκομένων, όπως γενικά στον τομέα των τεχνολογιών αυτών. Τέλος, πάνω από όλα, είναι απαραίτητη η τυποποίηση στο μέλλον να περιλαμβάνει την απόλυτη διαλειτουργικότητα. Πρέπει να έχουμε συστήματα τα οποία οδηγούν σε διαλειτουργικότητα σε συστημικό επίπεδο και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες της Ευρώπης τις υπηρεσίες που απαιτούν και να δώσουμε στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τη δυνατότητα να είναι οικονομικά επωφελής και επιτυχής. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς προτύπων θα πρέπει να σκεφτούν και περαιτέρω από την τωρινή κατάσταση και να μπορέσουν να εξεύουν τα εργαλεία που θα οδηγήσουν σε διαλειτουργικότητα. Χρειάζονται νέε ε, μέθοδοι δοκιμασία και πρωτοτυποποίηση και τρόποι κοινή οργάνωση στις ε, διαδικασίες βιομηχανικού χαρακτήρα και στη σημασιολογία και οντολογία που χρησιμοποιείται. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ενσωματωθούν στο γενετικό μας υλικό. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ για αυτή την σαφέστατη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Κατά τη διάρκεια της δικής μας συνάντησης σήμερα, η ICAN, οι φορείς του ίντερνετ, του διεθνού Διαδικτυακού συστήματο, συναντώνται σήμερα στι Βρυξέλλες. Και η ομάδα δράση για το διαδίκτυο συναντιόνται επίση και ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το τι θα συζητήσουμε σήμερα, συζητώντα για την διαλειτουργικότητα και άλλα τέτοια συστήματα. Θα υπάρξουν λοιπόν αντίγραφα που θα διατεθούν ε, εκτός αίθουσας από όλε τι παρουσιάσει. Με ιδιαίτερη χαρά μου τώρα να καλέσω τον κύριο Μπράιντε να μας μιλήσει. Τον άλλον τον ε, γνώρισα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητεία μας ε, τη Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς στη Γενέβη. Το 2004 νομίζω. Πάντως ε, βλέπω ότι το ενδιαφέρον του για, το, για τις προδιαγραφές εξακολουθεί. Εργάστηκε και στη Γαλλική, στο Γαλλικό Οργανισμό Τυποποίησης και άλλα είναι μεγάλη μας χαρά που θα μοιραστείς ε, μαζί μας την άποψή σου για τη στρατηγική θεώρηση του μέλλοντος της τυποποίησης. Έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κυρίες και κύριοι, μόλις έγραψε ένα άρθρο για ένα επιστημονικό περιοδικό με τον τίτλο «Τα πρότυπα φαίνονται βαρετά, ξανασκεφτείτε το. Την περασμένη δεκαετία τα πρότυπα έχουν ε, πάρει διαφορετική εικόνα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι εταίροι πρέπει να καλύψουν ε, διαφορετικές ε, απόψεις της, των προτύπων. Τη βιωσιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου να ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο φαίνεται εδώ και χρόνια να θεωρεί ότι τα πρότυπα δεν είναι βαρετά. Ίσα ίσα μπορούν να μας ανοίξουν δρόμους για το μέλλον. Εγώ τώρα με την πείρα που έχω την τελευταία δεκαετία και ήμουν προ, αντιπρόεδρος της ήμουν ταυτόχρονα και πρόεδρος της ε, έφνο. Οπότε θα ήθελα με την παρουσίασή μου να υπογραμμίσω τα εξής έχοντας μια σχετική ελευθερία έκφρασης. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα σημεία, τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες, τις απειλές για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να δείξω ποια είναι η σημερινή μας θέση και η δυναμική διάσταση των προτύπων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τυποποίησης. Πρώτα απ' όλα τα πλέον εκτήματα. Νομίζω ότι 20 χρόνια υλοποίησης της νέας προσέγγισης και η συνεχής αναφορά των ευρωπαϊκών προτύπων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ενισχύει ιδιαίτερα το δικό μας σύστημα τυποποίησης. Έτσι διασφαλίζεται η συμβολή των εταίρων πολυμερό τις τεχνικές λεπτομέρειες σχεδιασμού των οδηγιών και δεν είναι μια σταθερή βάση για την ανάληψη των ε, προτύπων από τις κυβερνήσεις και την αγορά. Βεβαίως, τα πρότυπα, τα υποχρεωτικά πρότυπα είναι το 30% της ε, παραγωγής της Ένσενελέκ, ενώ το 70% είναι εθελούσια πρότυπα. Βεβαίω κάποιε φορέ υπάρχει αντίφαση με τα εθνικά πρότυπα και το να αρθούν όλα αυτά όπω ήδη έχει να στην Ευρώπη είναι ένα από τα πλεονεκτήματά μα. Τώρα για την πολυμερή συνεργασία μα. έχει έρθει η στιγμή όπου η υλοποίηση της συμφωνίας του ΠΟΕ για τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο υποχρεώνει τις χώρες εκτός Ευρώπης να αναθεωρήσουν τα συστήματά τους τυποποίησης. Έτσι λοιπόν το ευρωπαϊκό μοντέλο ήρθε σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή. Επίσης, η Ευρώπη έχει κάποιους εθνικούς πρωταθλητές μεταξύ των εθνικών φορέων τυποποίησης. Δεν θα τους κατονομάσω. Αλλά υπάρχουν φορείς τυποποίησης στην Ευρώπη σε κάποια κρατη μέλη που διδραματίζουν πολύ ενεργό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο. Έτσι, οι συμφωνίες της Βιέννης και της Δρέσδης διασφαλίζουν την συμβατότητα με τη διεθνή πρότυπα και βεβαίως το πώς βαρύνουν η ISO, η IEC και η ITU στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερη σημασία εδώ. Τώρα ποιες είναι οι αδυναμίες. Νομίζω ότι η διατομιακή προσέγγιση στην τυποποίηση είναι μία από τις πρώτες αδυναμίες. Υπάρχει ένα παράδειγμα για ένα πρόγραμμα στην Ευρώπη όπου η σύγκληση των τεχνολογιών, οι διεπαφές που δημιουργούνται με το πολλαπλών πόλων σύστημα τυποποίησης δημιουργεί δυσκολίες. Να κάτι με το οποίο ασχολήθηκε λοιπόν η έτσι σε αυτό το σύστημα τηλεπικοινωνιών. Κάτι άλλο που αφορά πολλούς τομείς και που πρέπει να έχουμε διατομιακή προσέγγιση είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η τυποποίηση και πολλά περισσότερα νομίζω μπορούν να γίνουν εδώ. Είναι αμφίσιμη όμως η θέση της Ευρώπης σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να προωθούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε αντίθεση με τα αμερικανικά, λόγου χάρη. Ή να συνεισφέρουμε περισσότερο στο διεθνές σύστημα. Εκεί απαιτείται περισσότερη σαφήνεια. Επίσης το μοντέλο μας, παρά την πολυπλοκότητά του, είναι μονοδικό και οι τα, εργαλεία, των τα τεχνολογικά εργαλεία που στηρίζουν το σύστημά μας είναι καθοριστική σημασία. Τώρα, ποιοι είναι οι τομείς όπου περιμένουμε να έχουμε ευκαιρίε για να χρησιμοποιήσουμε νέα τεχνολογικά μέσα. Ε, τα, τα εθελούσια πρότυπα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αφορμές για να ενισχυθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνες. Επίσης, ε, χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, λόγου χάρη, είναι πολύ θετικό ότι συμμετέχουν στο διεθνές σύστημα, όπως κάνει και η Ευρώπη και ο ακαδημαϊκός χώρος είναι πολύ σημαντικό επίσης να συμμετέχει στην όλη προσπάθεια, όπως ε, συμβαίνει και με τα με τον σχεδιασμό των εργαλείων μας. Επίσης ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών θα καθορίσει το μέλλον των ευρωπαϊκών προτύπων. Όμως τα πρότυπα που στηρίζονται σε συμφωνίες για την ώρα επειδή έχουν διαμορφωθεί ανατομέα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Θα πρέπει λοιπόν στο διεθνέ σύστημα να υπάρξει με ένα συνδυασμό των ευρωπαϊκών με τα αμερικάνικα πρότυπα. Επίσης η εμπειρογνωμοσύνη που διατίθεται. Η ειδική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο να συνεργάζονται δεν είναι τόσο απλό σε δυσχερές ε, οικονομικό πλαίσιο. Μια επιπλέον απειλή είναι η ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου που έχει διαμορφωθεί για να στηρίξει την ευρωπαϊκή και εθνική τυποποίηση. Εδώ μπορεί να έχουμε παραβίαση των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την μείωση της ε, δημόσιας στήριξης, η ίδια χρηματοπιστωτική κρίση. Μπορεί να παράγει περισσότερους κανόνες και περισσότερη ανάγκη ρύθμισης σε αντίθεση με την ε, οικειοθελή τυποποίηση. Επίσης μπορεί να υπάρξουν τάσεις εθνικού προστατευτισμού λόγω της οικονομικής κρίσης. Τώρα, για τα εθνικά, <clears throat> για τα, για τα πρότυπα της Ευρώπης σε σχέση με τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης. Η θέση της Ευρώπης είναι σταθερή, με μια ελαφρά διάβρωση να παρουσιάζεται σε κάποια επίπεδα επιτροπών και κυβερνήσεων. Έχουμε 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, ΆΙΖΟ σε κάθε περίπτωση. Και τώρα ορισμένε συστάσεις συστήνω η νέα προσέγγιση να καλύψει και άλλους τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών και των ζητημάτων αηφορίας. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω παρά να αποσταθεροποιηθεί. Επίσης, νομοθετικές αποφάσεις θα, θα, θα χρειαστούν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής θέσης στο διεθνές σύστημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλαν, ήταν πάρα πολύ νοπή και ενδιαφέρουσα αυτή η προσωπική σου παρουσίαση και νομίζω ότι μπορείς να παίξεις ένα ρόλο όπως αυτό που παίζει ο πρόεδρος ο κ. Μόντι για τον πρόεδρο Μπαρόσο, δηλαδή να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργειών στον τομέα αυτό. Πολύ χρήσιμο είναι αυτό λοιπόν και χαίρομαι που αναφερθήκατε ιδιαίτερα για ορισμένα από τα θέματα τα οποία συνάπτονται με τη βιωσιμότητα. Ιδίω με τη βιωσιμότητα. Ακούσαμε για τις δημόσιες προμήθειες προηγουμένως, γιατί η Επιτροπή μας έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην έκθεσή της, της κυρίας Ρούλε για τις δημόσιες προμήθειες. Και εκεί αναφερθήκαμε στις, στα πρότυπα. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό με έναν τρόπο ο οποίο είναι συνεκτικός. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό τον γύρο. Δίνω το λόγο στον κύριο Μακ Λόου, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Βρετανικού Ιδρύματος για τα πρότυπα. Ιδιαίτερα ενεργός ήταν πάντα ο κύριος Λόγου για τα θέματα αυτά και έχει φτάσει στα πρότυπα μετά από μια διακεκριμένη καριέρα στην βιομηχανία και επομένω σίγουρα γνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα πρότυπα και πιστεύω ότι θα μπορέσει να το κάνει και τώρα. σα δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Εκπροσωπώ την ε, έκθεση του πάνελ των ειδικών. Βεβαίως ε, δεν μπορώ να τα παρουσιάσω όλα αυτά στον χρόνο που μου δίνετε, οπότε ελπίζω τουλάχιστον να δείτε τη σύνοψη αυτής της έκθεσης σας. Δεν παρακαλώ την πρώτη διαφάνεια. Να. Συνεχίζω κύριε Πρόεδρε. Το πάνελ αυτό, το λεγόμενο Express, αποτελείται από 30 ειδικού ε, και συνεδρίες τον Ιανουάριο φέτος υπάρχουν 12 ε, στόχοι και 30 συστάσεις. Θα αναφερθούμε λίγο στους ε, στόχους αυτούς. Επίσης βλέπετε πως τα έχω κάνει εδώ πέρα, τα έχω κωδικοποιήσει με χρώματα, Τέλο πάντων με τα χρώματα του Βρετανικού φαναριού, όχι τα τυποποιημένα. Βλέπετε πως ε, έχουμε εδώ πέρα τα κράτη-μέλη του ΆΙΖΟ και τη Κομισιόν. Τι βλέπουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ε, βλέπουμε πως ένα σύστημα ισχυρό και αποτελεσματικό και με τους τρεις ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης, ε, συνεισφέροντας έτσι και στις ανάγκες κοινωνίας των επιχειρήσεων και της ε, πολιτικής. Βλέπουμε λοιπόν πως έχουμε μεγάλη διεθνή επιρροή, έχουμε άνω από το 50% του δουσού του ΑΕΖΟ και μεγαλύτερη προσώπηση στις επιτροπές από όσο είναι η οικονομίες και οι περισσότερες προδιαγραφές ε, παγκοσμίω προέκυψαν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Έχουμε λοιπόν μια επιτυχία η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Επίσης είμαστε πολύ καλά προσανατολισμένοι στην αγορά, ειδικά σε εθνικό επίπεδο και συμμετοχή στην καινοτομία. Αν δείτε τις μελέτες για τα οικονομικά ωφέλη θα δείτε πως ε, η διασφορά της ε, καινοτομίας γίνεται κυρίως μέσω των προδιαγραφών. Η οικονομική συνεισφορά της διαδικασίας είναι πολύ μεγαλύτερη από το επίπεδο χρηματοδότησης και της Κομισιόν και των κρατών μελών κατά τάξης μεγέθους. Επιβεβαιώνουμε τα συμπεράσματα της Κομισιόν στο έγγραφο του 2008 που νομίζω αποτελούσαν μια πάρα πολύ καλή βάση για να διατηρηθεί αυτή η απόδοση και να βελτιωθεί. Βρήκαμε όμως κάποιους τομείς ε, οι οποίοι ήδη αναφέρθηκαν, στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε. Πρέπει να επεκτείνουμε να επεκταθούμε στον τομέα των υπηρεσιών στην Ευρώπη που είναι κυρίαρχος. Πρέπει επίσης να, είναι, να γίνουν γνωστά τα ωφέλη των προδιαγραφών. Ίσως να είναι κάτι το βαρετό, αλλά συχνά είναι κάτι το άγνωστο. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ομάδων εκείνων, ειδικά των ομάδων με αναπηρίες που μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες προδιαγραφών και να δούμε το ζήτημα του κόστους κύκλου ζωής. Πρέπει επίσης να εμπλακούμε νωρίτερα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για να συνεισφέρουμε και με τις ανάγκες της αγοράς με τρόπο συνεκτικό. Πρέπει να εμπλακούμε στα προγράμματα έρευνα της Κομισιόν και να αποτελέσουμε μέρος των προτεραιοτήτων που δίνονται αν είναι να είμαστε να έχουμε διεθνή ηγετικό ρόλο. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που έχουμε θετικό, την ανοτεχνολογία. Πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των ατύπων εκείνων φορέων. Δεν θέλω τώρα ε, να τα λέω εγώ κονσόρτσια ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν εξαιρετικούς μηχανισμούς για να έχουν καλύτερες ε, διαδικασίες για να δούμε ακριβώς ε, πώς θα ενσωματωθούν στην άσκηση της πολιτικής. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί η εμπλοκή και η ενεργό συμμετοχή του τομέα της εκπαίδευσης επίσης και εκεί πέρα νομίζω κάποια έχουν κάποιες καλές πρακτικές οι οποίες όμως πρέπει να επεκταθούν. Τώρα θα αναφέρω τους στόχους γρήγορα. Στόχος 1, ανταγωνιστικότητα, όπως ακούσαμε, σε διεθνές επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το υψηλό επίπεδο επιρροής και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ε, το τι σημαίνει αυτό παγκοσμίω. Ειδικά οι Κινέζοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το τι κάνουμε, ε, πώ θα κάνουμε τα πράγματα στην Ευρώπη. Επίση, όσον αφορά την καινοτομία, πρέπει να περάσουμε το μήνυμα πω οι φοροδιαγραφέ ε, μεταφέρουν την καινοτομία στην αγορά. Στόχο 3 και 4. Συνεκτική προσέγγιση να συνεργαστούμε με την Κομισιόν και τις διάφορες γενικές διευθύνσεις στο τομείς έρευνας και της εκπαίδευσης. Δεν υπήρχε σύνδεση στο παρελθόν και μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα για να επηρεάσουμε τους ηγέτες ε, του μέλλοντος. Στόχος 6 τομέας των υπηρεσιών προφανώς να υπάρξει μια τυποποίηση στις υπηρεσίες που δεν υπήρχε στο παρελθόν, αλλά βεβαίως να μην ε, πνίξουμε τον τομέα, πρέπει να το δούμε ανά περίπτωση. Στόχος 8, να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα τυποποίησης ε, μία προφανής εξέλιξη από τη δουλειά την οποία κάνουμε. Χαιρόμαστε που βλέπουμε την ε, ΣΕΝ και την ΕΛΕΚ και την AGM που συνεργάζονται για να δουν τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον. Και οι πρόσφατες αλλαγέ στην ΕΝΕΛΕΚ αποτελούν απόδειξη ότι πράγματι έχουμε αλλαγές. Στόχος 9 τα διάφορα φόρα και κοινοπραξίε. Όπω είπαμε, υπάρχει μεγάλη συνεισφορά όχι μόνο στον τομέα τηλεπικοινωνιών και πληροφορική και άλλοι τομεί όπω η υγεία που πρέπει να μας απασχολήσουν για το περιεχόμενο παράγεται εκεί πέρα. Και πρέπει να ε, το εξετάσουμε και αυτό, αλλά βέβαια δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τις κοινοπραξίες απομονωμένες. Ε, η έκθεση Express συνιστά ένα γενικότερο ε, σχέδιο δραστηριότητας για να ε, συνεργάζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι στον αφορά και όσο πιο γρήγορα το κάνουμε τόσο το καλύτερο στόχος 10 πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα υπάρχει ένα έργο α, που κάνει η ΣΑΝ και η ΣΑΝ για καλύτερη πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά λοιπόν την τιμή, πρόσβαση, εμπλοκή, επιρροή και πάρα πολλές καλές πράκτικες που χαίρομαι που τις βλέπω. Στόχος 11 χρηματοδότηση όπως είναι προφανές σε καιρούς ύφεσης ε, πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα χρήματά μας. Η έκθεση Τεχνόπολης ε, που παρέγγειλε η Κομισιόν αποτελεί εξαιρετική βάση για να δούμε πώς θα επενδύσουμε στη διαδικασία τυποποίησης και τέλος στόχος 12 το νομικό πλαίσιο νομίζω πως πρέπει εδώ πέρα να δώσουμε δυνατότητα να γίνουν οι βελτιώσεις που θέμε και να μην τις εμποδίσουμε. Να καταλήξω τώρα, πιστεύω πως είμαστε σε πολύ καλή θέση για να έχουμε μια ισχυρή βάση για το 2020. Έχουμε μια σειρά βελτιώσεων που μπορεί να γίνουν και κατά βάση είναι η ανάγκη να υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο σε ολόκληρη την Ευρώπη για να συνεχίσουμε να έχουμε διεθνή επιρροή όπως ε, έχουμε και αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την προσέγγιση των ESO αυτή τη στιγμή για τις διαδικασίες τους και θα πρέπει να αρχίσουμε να μέναμε πολύ περισσότερο για τα ωφέλη της τυποποίησης. Τελευταία τελευταία διαφάνεια παρακαλώ. Λοιπόν, το ευρωπαϊκό σύστημα του 2020 τι μορφή πρέπει να έχει. Πρέπει να είναι ακέραιο να προσφέρει ωφέλη στην κοινωνιακές επιχειρήσεις και σε όλες τις πτυχές ε, των αναγκών του καταναλωτή. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό να αφορά το κόστος, να αντικατοπτρίζει ισορροπημένα τους στόχους ε, της ε, πολιτικής και βεβαίως αποτελεί υποκατάστατο για την ρύθμιση και βεβαίως θα επιφέρει και συνεχή βελτίωση για να διασφαλίσουμε πως ε, θα έχουμε καλύτερες προοπτικές σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε η Κομισιόν στην αναθεώρηση την οποία θα κάνει θα πρέπει να δει αυτές τις βελτιώσεις για να ενισχύσει τα ισχυρά μας σημεία και να ενθαρρύνει τα στοιχεία εκείνα που θέλουμε για να προχωρήσουμε προς το 2020. Ευχαριστώ. Uh, well, thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόου και όλη την ομάδα σας η οποία έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να μας δώσει αυτά τα ενάρσματα στη συζήτησή μας. Έχουμε τώρα περίπου 20 λεπτά για συζητήσεις με τα από τα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής μας θα προσκαλέσω τον εισηγητή για να θέσει πρώτα ερωτήματα και θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής μας να είναι σύντομοι και συνοπτικοί ώστε να μπορούν τα μέλη του πάνελ να απαντήσουν με πλήρη τρόπο. Κύριε και η κυρία Κόνη η οποία είναι η σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ, δεν ξέρω για τους σοσιαλιστές οι υπόλοιποι και οι υπόλοιποι θέλουν να λάβουν το λόγο κυρία Βάλλη Σαντομόζα. Λοιπόν, ίσως ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα. Μπορείτε λοιπόν να δώσετε περίπου ένα λεπτό σε κάθε ερώτημα, ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο για να απαντήσουν τα μέλη του Πανεπιστημίου Βοζασικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονές μας. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμε οι παρουσιάσει του και έχω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω για τον Κέβιν. Συναντηθήκαμε στη Γενέβη και προσωπικά μπορώ να πω ότι το ταξίδι μας στη Γενέβη ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Συναντηθήκαμε με διεθνείς οργανισμούς και ο Κέβιν αναφέρθηκε στην παρουσία του το γεγονός αυτό και ο κ. Μπράιντεν επίσης. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Είναι καλύτερο να είναι η Ευρώπη εκπροσωπούμενη από 27 συν 4 φορεί σε επίπεδο ψήφων. Πιστεύετε με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τις κοινέ μας πολιτικές ή μήπως είναι καλύτερα να έχουμε ένα ή δύο μονάχα άτομα τα οποία εκπροσωπούν συνολικά την Ευρώπη στις συζητήσεις του, των διεθνών φορέων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο Λόου υπεύθυνο του πάνελ για την αναθεώρηση. Γιατί από μια άποψη φαίνεται ότι το σύστημα της τυποποίησης σήμερα δείχνει ότι το πρόβλημα είναι η πρόσβαση και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων εταίρων στην όλη διαδικασία ισότιμα. Ιδίω αυτό παρουσιάζει δυσκολίε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβαση και συμμετοχή, γιατί αυτό θα επέτρεπε να ωφεληθεί και το ευρωπαϊκό σύστημα της αγοράς και βέβαια και το διεθνές. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το σύστημα και ως προς την ε, δομή του, τη διάρθρωση δηλαδή των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων και της εκπροσώπησης όλων των φορέων που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα. Uh, thank you very much, Mr. Όχι. Θα ήθελα να τονίσω ότι εγώ έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν τα ζητήματα τυποποίησης. Είχα θέσει το ερώτημα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με καλύτερο τρόπο τα υποδείγματα τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρξει πραγματικά μια εγγύηση ότι τα πρότυπά μας θα οδηγήσουν και σε καλύτερη παραγωγή προϊόντων. Ελέγχθη προηγουμένως ότι τα πρότυπα και η προτυποποίηση είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και της έρευνας και της καινοτομίας. Προφανώς θα πρέπει όμως να δούμε καλύτερα ποια είναι η σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας, μεταξύ έρευνας και παραγωγής. Η πραγματικότητα μπορεί πράγματι να εμπλουτίσει και τη θεωρία. Θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποιες πρόσθετες πληροφορίες από σας. για το τρόπο με τον οποίο εμεί μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, τυποποίηση. Uh, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ, Λεωπρόδος θα ήθελα να εκφράσω. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πληροφορικά αυτά τα οποία ακούσαμε. Έχω δύο ερωτήσεις. Μιλάμε για την τυποποίηση των υπηρεσιών. Έχω το ερώτημα εάν θεωρείτε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια νομική βάση για τις υπηρεσίες και για τα αγαθά. Γιατί έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί υπάρχουν κάποιες ε, ιδιαιτερότητε. Δεν ξέρω αν λοιπόν θεωρείτε ότι επαρκεί μία νομική βάση ή αν θα πρέπει να γίνει μία διαφοροποίηση, ειδικά όσον αφορά την υγεία. Και το άλλο ερώτημα αφορά την πρόσβαση. Οι συνθήκες στα κράτη-μέλη διαφέρουν. Υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία πραγματικά η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το συνδέσμο καταναλωτών, περιβαλλοντικών ενώσεων ε, είναι διασφαλισμένη. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν κάτι μέλη τα οποία δεν λειτουργεί τόσο καλά. Και αν αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσουμε να το ισχύσουμε αυτό, γιατί δεν ξέρω κατά πόσον είναι σωστές οι εθνικές αντιπροσωπείες, αλλά δεν είναι όλες ίδιες και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να φροντίσουμε για περισσότερη διαφάνεια. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Βάιλερ. Ευχαριστώ και από μένα. Συμφωνώ αυτά τα οποία είπαν οι ειδικοί συχνά υποτιμάμε τη σημασία των προδιαγραφών συχνά μόνο όσοι δουλεύουν πάνω στο αντικείμενο αντιλαμβάνονται το πόσο βοηθάει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο από την βιομηχανία. Δεν γίνεται στο κενό αυτή η συζήτηση, αναφέρεται στα σχέδια της Κομισιόν για νέες προτάσεις που θα υποβάλει το φθινόπωρο και υπάρχει ήδη μια ανάλυση της ε, Κομισιόν για το ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν αρκετά, δεν επωφελούνται αρκετά, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε τυποποίηση και προδιαγραφές όπως θα έπρεπε και αποτελεί βεβαίω επίση η τυποποίηση και τη νομοθεσία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Οπότε το ερώτημα μου είναι τι μπορούμε να κάνουμε από ευρωπαϊκή πλευρά για να συμμετέχουν καλύτερα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να μην είναι πολύ υψηλό το κόστο. Νομίζω πω όλοι πλην ε, Λουξεμβούργου πρέπει να, παντού πρέπει να πληρώνουν. Γιατί δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι υπόθεση των μεγάλων επιχειρήσεων. Uh, Ευχαριστούμε κυρία Σαλδεμόζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν έχω γραβάτα για να σας δείξω τι έχουμε καταφέρει στους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης. Όμως το μήνυμα θα πρέπει να περάσει προς τους καταναλωτές. Είναι σημαντικά τα πρότυπα. Και εγώ έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Λέτε ότι είναι σημαντικό να φτάσουμε σε τυποποίηση και στον τομέα των υπηρεσιών. Θα ήθελα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ποιε είναι οι υπηρεσίε ε, που έχετε υπόψη, Πού χρειάζονται περισσότερα πρότυπα και προδιαγραφέ. Καταλαβαίνω ότι εννοείται με την τυποποίηση για τα προϊόντα τηλεπικοινωνιών, τα τεχνολογικά, αλλά για τι υπηρεσίε θα ήθελα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ευχαριστώ. Um, um, Και τέλος, η σκληρά εργαζόμενη πρόεδρός μας, αντιπρόεδρός μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για την ποιότητα των παρέμβασεων τους. Το ερώτημά μου απευθύνεται προς όλους, βεβαίως, αλλά κατεξοχήν προς τον κύριο Φίλιπς. Είπατε κάτι που πραγματικά μου άρεσε ιδιαίτερα. Νομίζω η Ευρώπη έχει μια κραυγαλαία αδυναμία εδώ. Είπατε ότι πρέπει να χτίσουμε το κοινοτικό ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν αφορά μια πολύ σύγχρονη και πολύ μεγάλη πρόκληση. Και σε σχέση με τα ερωτήματα που τέθηκαν, έχω και εγώ ένα ερώτημα. Για την ε, κατανομή του κόστους. Δεν θεωρείτε ότι θα ήταν ε, μεγάλη και σημασία να γίνει μια σοβαρή εκστρατεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Μαζί και οι πολιτικοί ηθήνοντε και οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οι ενώσει καταναλωτών και οι ερευνητέ σε σχέση με την καινοτομία. Και όλα αυτά να περάσουν και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα που δεν έχει καθόλου ενημέρωση, καθόλου πληροφορίες για όλα αυτά. Αυτά είναι, αυτό είναι το δικό μου ερώτημα για το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Και θα σας ευχαριστούσα να αναπαντούσετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ και τώρα θα καλέσω τους ομιλητές από το πάνελ μας να απαντήσουν. Θα σας δώσω περίπου ένα λεπτό στον καθένα. Όμως, για κάποια τα ερωτήματα που τέθηκαν, ότως ή άλλως θα ακούσουμε και άλλους ομιλητές αργότερα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία. Ο Κέβιν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι ένα από τα ερωτήματα τα οποία απευθύνονται άμεσα σε μένα αφορούσαν ένα υποθετικό και προκλητικό σενάριο κατά κάποιο τρόπο να περάσουμε από 27 ψήφους για την Ευρώπη σε μία μοναχα ψήφο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι υποθετικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το εξετάσουμε. Νομίζω ότι η διαδικασία του ISO βασίζεται στη λειτουργία ενός συστήματος. Κάθε χώρα έχει μία ψήφο. Αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Και η ISO και η ISC λειτουργεί έτσι. Η διαδικασία στους φορείς μας επίσης βασίζεται σε μία σύνδεση με τους εθνικούς φορείς, με τους εμπειρογνώμονες, με τους εκπροσώπους των χωρών αυτών που είναι εκπρόσωποι συγκεκριμένων χωρών και των απόψεών τους. Τρίτον, η συμφωνία της Βιέννης και της Δρέσδης με την ΑΕΣΥ, με τη Σένελεκ, αυτές βασίζονται στην ιδέα αυτή ότι κάθε χώρα έχει μία ψήφο. Επομένως, αν αναθεωρηθεί αυτό, πρέπει να ξαναδούμε και αυτές τις συμφωνίες. Η Έλενα Σαντιάγου. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω για την ερώτησή σας ε, για την πρόσβαση και για κάποιε από τι ερωτήσει των βουλευτών να απαντήσω τα εξή. Η Sensa NL ξεκίνησε μια μελέτη πριν από τριετία. Έχουμε δώσει 58 συστάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ε, τυποποίηση. Έχω λοιπόν μια πρώτη και άμεση απάντηση γιατί με το νόμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Small Business Act, Act ε, στην, στο τοπό μας συμπεριλάβαμε όλα τα δεδομένα και όσα λείπουν θα δημοσιευτούν ως το τέλος της χρονιάς. Τα μέλη μας κάνουν ακριβώς το ίδιο στο δικού τους εθνικούς ιστοτόπους, στη γλώσσα τους. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Αυτό που είναι ιδιαίτερη σημασία είναι ο ρόλος που διδραματίζουν οι εθνικοί οργανισμοί και οι εθνικοί φορείς τυποποίησης. Διότι μπορεί να αληθεύει ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν ακόμη επισήμως στις, ε, στους ευρωπαϊκούς φορούς αλλά το κάνουν μέσω των τομεακών τους οργανώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις επενδύσεις και τις προσπάθειες εκπαίδευση και την υποστήριξη από τα κάτι μέλη προς τους εθνικές εγκαλιστικές οργανώσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι καλύπτονται όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα και ενημερώνονται. Και όλοι μας βοηθούν πάρα πολύ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, συμμετέχοντας και θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα. Έχουμε και ένα helpdesk, ένα γραφείο υποστήριξη, το οποίο είναι ελεύθερο στην πρόσβασή του, Βρίσκεται, μπορεί κανεί να έχει πρόσβαση και μέσα στο τόπο. Οπότε, όποιο θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μα, με το δίκτυό μα και τα εθνικά μα μέλη, μπορεί να το κάνει. Οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση από μια ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να απευθυνθεί σε έναν εθνικό φορέα τυποποίηση και στη δική του χώρα. Βεβαίω πολλά απομένουν ακόμη να γίνουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και αυτό θα μα ωφελήσει όλου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φίλιπς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου τέθηκε το ερώτημα για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινότητες ενδιαφέροντος γύρω από την τυποποίηση. Ιδίω στην Ευρώπη, διασφαλίζοντα την οικονομική επιτυχία της τυποποίησης. Το πρώτο βήμα για να γίνει βεβαίως αυτό είναι να εντοπίσουμε τους στόχους μας, δηλαδή μια δράση για να ορίσουμε στόχους. Παραδείγματα επιτυχίας. Όταν χτίσαμε το πρόγραμμα εταιρική σχέση τρίτη Γενιά, στην ΕΤΣΙ, είδαμε ότι το πρόγραμμα αυτό είχε επιτυχίε σε όλο τον κόσμο. Ένα παράδειγμα αποτυχία βεβαίω είναι αυτό της ασύρματης πρόσβασης στο ίντερνετ. Εκεί έτσι είχε ένα προϊόν, ε, το Highland, το οποίο ήταν ε, πολύ υψηλή τεχνολογικής, ε, ήταν προηγμένης τεχνολογικής κατασκευής, αλλά τελικά δεν πέρασε γιατί δεν είχε κάποια τεχνικά προβλήματα. Τελικά επικράτησε το πρότυπο 802.11. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να χτίσουμε αυτές τις κοινότητες ενδιαφερόντων και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσοι δρούν στον οικονομικό τομέα και οι ενώσει του, οι οργανώσει του, θα δημιουργήσουν τι πρώτε κοινότητε οικονομικού ενδιαφέροντο. Αυτό νομίζω ακριβώ λείπει σήμερα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ευχαριστώ. Alan Δράτω με τις ευκαιρίες να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις, εκτός μικροφώνου κύριος Μπράιντεν. Το πρώτο είναι τι θα συνέβαινε αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μία έδρα αντί για 27. Συμπληρώνοντας τον συνάδελφο, θα πω πως θα υπήρχε και σοβαρό νομικό πρόβλημα για τον Άιζο, γιατί βασίζεται σε εθνικό σε εθνική συμμετοχή και όταν ξεκινάει κανεί την επανάσταση βεβαίω, ξέρει πω ξεκινά αλλά δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Δεύτερο σχόλιο για τι υπηρεσίε Ο Άιζο. Η δραστηριοποιείται ήδη σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν τομεί όπω οι υπηρεσίε υδάτων, ο τουρισμό πληροφορική ε, που, ανα... που ήδη απασχολούν τον Άιζο. Οπότε η έννοια της ε, προσέγγισης αυτής πολλών συμμετεχόντων ε, με βάση τη συνένεση για την ε, ποιότητα και την περιοχή των υπηρεσιών ήδη υπάρχει. Ευχαριστώ και τέλος Mike Λόου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες. Και άλλοι, π.χ. οι μειονότητες, πώς μπορούν να εμπλακούν στις ε, προδιαγραφές. Αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση, γιατί είναι δύσκολο βέβαια να είναι κανείς όντως παρόν, αλλά ε, ήδη υπήρχε κάποια ε, πρωτοπορία και τώρα εξαπλώνεται. Είναι η εμπλοκή μέσω διαδικτύου στην ανάπτυξη των ε, προδιαγραφών. Έχουμε συμμετοχή πάνω από 10.000 μικρών φορέων ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο που ανέπτυξαν προδιαγραφές ε, και συμμετείχαν. Το επόμενο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το μέσο των υπηρεσιών. Όπως είπε ο Άλλαν και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλές τέτοιες προδιαγραφέ για τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται. Εγώ θα αναφέρω την έκθεση της Κομισιόν που ανέφερε την ανάγκη τυποποίησης των υπηρεσιών, αλλά πρέπει βεβαίως αυτό να γίνει από την αγορά. Ο τομέας των υπηρεσιών πρέπει να μας πει πού θέλει τυποποίηση και όχι η πολιτική ή κάποιοι φορείς προδιαγραφών να τους εξαναγκάσουν. Και η έκθεση το αναφέρει αυτό και το αντιμετωπίζει αρκετά καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα γίνει ε, συζήτηση, θα ακούσουμε την κυρία Βλάχα αργότερα, για τις υπηρεσίες, οπότε προτείνω να ακούσουμε τότε και αυτά τα οποία θα πει η κυρία Σχαλντεμόζε. Και νομίζω έγινε και μια καλή εισαγωγή. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, πάρα πολύ. Νομίζω πως πρέπει να χειροκροτήσουμε το πρώτο μας πάνελ. Ήσασταν ε, φανταστικοί. Uh, και τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα της ακροασής μας για την τυποποίηση ως υποστήριξη κοινωνικών και δημοσίων συμφερόντων. Συζητήσαμε ήδη το θέμα της συμμετοχής της κοινωνίας στην εξέλιξη των προτύπων και χαίρομαι με μεγάλη, έχω μεγάλη χαρά, μπορώ να χαιρετήσω την παρουσία του κ. Στίβεν Ράσελ, του Γενικού Γραμματέα της ΑΝΕΚ, που θα μας πει πώς θα ενισχύσουμε τη φωνή του καταναλωτή στην ανάπτυξη των προτύπων, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, με τα flotters από την οργάνωση πολιτών για τα πρότυπα σε επίπεδο περιβάλλοντος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως τα πρότυπα του περιβάλλοντος είναι υψής της σημασίας για το έργο μας, και ο Στέφανος Μπόι, ο, ο είναι ε, στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ε, εργατικών ενώσεων σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια για την προώθηση των προτύπων στους τομείς αυτούς. Επτά λεπτά θα έχει ο καθένας. Πάλι θα πρέπει να είμαι αυστηρός για να μπορούν όλοι να έχουν το χρόνο που χρειάζεται και να υπάρξει και συζήτηση. Έχουν 7 λεπτά λοιπόν ο καθένας. Ξεκινώ με τον Στίβεν Ράσελ και σας δίνω με μεγάλη χαρά το λόγο σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Η ενιαία αγορά επιτρέψει στους καταναλωτές να αποφεληθούν από μια ευρύτερη επιλογή προϊόντων δεν χωρεί αμφιβολία ότι αυτή η προσέγγιση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αλλά η ενίσχυση αυτής της ε, διαδικασίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υφίστανται. Το θέμα της συνρύθμισης όπου υπάρχει η παρουσία των ε, εμπλεκομένων στην αγορά μέσα από φορείς όπως το έτσι και συγχρόνως η νομοθετική διαδικασία θα πρέπει κάπως να συνενώνονται. Η προτυποποίηση όπως βλέπετε είναι μια ουσιαστικά ιδιωτική υπόθεση. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ληφθεί το δημόσιο συμφέρον υπόψη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Και αυτό κάνει πολύ δύσκολο να υπάρχει μια διτή διαδικασία ρύθμισης που περιλαμβάνει και νομοθετικά μέτρα. Για να μπορέσει η τυποποίηση να οδηγήσει σε κάλυψη των αναγκών νομοθετικής ρύθμισης, όπως είπαν και ορισμένοι, τότε θα πρέπει οι δημόσιοι φορείς να εξασφαλίσουν ότι λαμβάνεται υπόψη και το δημόσιο συμφέρον σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά η ανάπτυξη των προτύπων είναι μια ανοιχτή διαδικασία καταρχήν, αλλά οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες κερδίζουν περισσότερο από την, από τον επηρεά, από την επιρροή τους σε αυτή τη διαδικασία και είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την εμπειρογνωμοσύνη για να συμμετάσχουν σε τέτοιους φορείς προτυποποίησης. Αντίθετα, οι καταναλωτές δεν έχουν την απαραίτητη πείρα και γνώση ή πολλές φορές είναι ανύπαρκτη η γνώση από την πλευρά των καταναλωτών σε πολλές χώρες. Η, πρό, ε, η μελέτη αυτή μάλλον για την πρόσβαση στην προτυποποίηση είδε ότι μόνο οριακά εκπροσωπούνται οι οργανώσεις των καταναλωτών σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη θεσμοποίηση τη συμμετοχή των καταναλωτών, όπω έχει γίνει και με την ΑΝΕΚ από το 1995. Επίσης, όπως λέει και η έκθεσή μας, η ΑΝΕΚ υποστηρίζει το σύστημα των εθνικών αντιπροσωπιών στη ΣΕΝ και ΣΕΝΕΛΕΚ, εξασφαλίζοντας ότι και η φωνή μια από τις πιο ασθενικές ομάδες συμφερόντων των καταναλωτών ακούγεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θέλω να θίξω την έτσι, Τζον, τα πρώτη της όπω το GSM έχουν βοηθήσει πάρα πολύ του καταναλωτέ και η ΣΕΝ και η ΣΝΕΛΕΚ με τα πρότυπά τους έχουν αντιμετωπίσει πολλά θέματα που ενδιαφέρουν του καταναλωτέ. Αλλά η παρουσία των καταναλωτών δεν είναι μονάχα το να εξηγούμε σε εθελοντέ καταναλωτέ ποιοι είναι οι κανόνε του παιχνιδιού. Θα πρέπει οι εθελοντές αυτοί από τους καταναλωτές να είναι και εμπειρογνώμονες στα θέματα για τα οποία συμμετέχουν στις συνεδριάσεις. Ας δούμε παραγωγικά το θέμα της ασφάλειας των παιδικών παιχνιδιών. Υπάρχουν 31 χώρες που συμμετέχουν και η ΑΝΕΚ έχει 6 εμπειρογνώμονες που έχουν αρκετή εμπειρογνωμοσύνη για να είναι σημαντικοί, έχουν σημαντικό λόγο σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα των καταναλωτών για την προστασία <clears throat> της ασφάλειας των καταναλωτών. Χωρίς την ΑΝΕΚ λοιπόν, μόνο 6 από τις εθνικές αντιπροσωπείες θα μπορούσαν να έχουν εμπειρογνωμοσύνη σε επίπεδο καταναλωτών και τι θα γινόταν στην περίπτωση των καταναλωτών στις υπόλοιπες 25 χώρες όπου δεν, έχει καμία, δεν υπάρχει καμία γνωμοδότηση από την πλευρά εμπειρογνωμόνων ε, για τα θέματα του καταναλωτή. Θα ήταν λοιπόν ανύπαρκτη ή ελάχιστη η συμμετοχή των καταναλωτών. Επομένως, χωρίς την ΑΝΕΚ δεν μπορεί να υπάρξει η εκπροσώπηση των καταναλωτών και είναι απαραίτητο να υπάρξει δημόσια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πρότυπα τα οποία είναι προ το καλό όλων στην κοινωνία και όχι μονάχα των λίγων εκλεκτών. Δυστυχώ. Αυτή η χρηματοδότηση δεν έχει αυτή τη στιγμή νομική βάση. Η χρηματοδότηση τη ΑΝΕΚ που είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ είναι τμήμα ενός προγράμματος για τους καταναλωτές που αποφασίζεται κάθε λίγα χρόνια από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Το 2013 εκπνέει αυτό το πρόγραμμα και ακόμα και αν υπάρξει ένα περαιτέρω πρόγραμμα δεν ξέρουμε αν ο προπολογισμό θα είναι επαρκή για να υποστηρίξει την ΑΝΕΚ, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλε απαιτήσει από τον προπολογισμό τη Γενική Διεύθυνση Υγεία και Καταναλωτών. Η ΑΝΕΚ λοιπόν προτείνει να υπάρξει και μια εγγύηση για την εκπροσώπηση των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θέλουμε τώρα να δούμε σε επίπεδο δομής να υπάρξει κάποια ριζική αλλαγή. Κυρίως δεν θέλουμε να δούμε μια περαιτέρω κατακαιρμάτιση, ένα κατακαιρματισμό του ευρωπαϊκού τομέα τυποποίησης πέραν τη ΣΕΝ, και έτσι. Δεν θέλουμε να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός φορέας τυποποίησης, γιατί δεν έχει νόημα να αποσυνδέσουμε την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων από διεθνείς και εθνικές δραστηριότητες, ούτε να οδηγηθούμε σε ένα διαχωρισμό σε, σε διάφορους φορείς. Κάποια τμήματα του έργου στην τυποποίηση ενδιαφέρει τους καταναλωτές, αλλά όχι όλα. Αν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πιστεύουν ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίηση πρέπει να παρέχει ακόμα περισσότερες εγγυήσεις σε μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά της ε, νομοθεσίας, η ΑΝΕΚ θεωρεί ότι αυτές οι εγγύησεις θα πρέπει να παρασχεθούν μέσα στο τωρινό σύστημα. Θα ήταν καλύτερο την Κομισιόν να συνεργάζεται με την ΕΤΣΙ, την ΣΕΝ και την ΣΕΝΛΕΚ για να υπάρχει και δεύτερος, μια δεύτερη γραμμή παραγωγής προτύπων σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον καταναλωτών. Υπάρχει ήδη το σύστημα αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα σύστημα για, που να περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους, όπως παραδείγματος χάρη στο στάνταρ 26.000 της ISO για τη συμμετοχή των εμπλεκομένων και είναι απαραίτητο να παραμείνουν οι εθνικές διασφαλίσεις με το να συμμετέχουν οι εθνικοί φορείς και να υπάρχει η δυνατότητα τα ευρωπαϊκά στάνταρ να γίνονται και εθνικά στάνταρ. Το να έχουμε μια προσέγγιση υπέρ των εμπλεκομένων ή μια διαδικασία μόνο εθνικών ε, οργάνων θα μπορούσε να γίνει δεκτή βάση της οδηγίας 98-34. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσει όπου έχει αποτύχει το παραδοσιακό σύστημα, ιδίως στην περίπτωση να υπάρχει ένα στάνταρ για τις ε, σκάλες στα σπίτια που χρειάστηκε 10 χρόνια για να ευδοκιμήσει. Εν κατακλείδη, είναι σημαντική τυποποίηση για την ε, ενία αγορά, αλλά εξακολουθεί να είναι μια ιδιωτική διαδικασία και αν πρόκειται να αντικαταστήσει την νομοθεσία θα πρέπει να περιλάβει και τους πιο αδύναμους και ανύπαρκτους εμπλεκομένους σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Στίβεν, για αυτές τις πολύ χαρακτηριστικές και υποδειγματικές συστάσεις προς την Επιτροπή μας. Ο κύριος Λότες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριοι βουλευτές, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη φωνή τη οίκο της ε, δική μα οργάνωση, περιβαλλοντική οργάνωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τους, ε, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις περιβαλλοντικές, ε, Είμαστε μη κερδοσκοπή οργάνωση και έχουμε 21 μέλη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατά μέλη του Όπως ξέρετε, μέλη είναι ενδεχομένως η ΒΒΕΦ, οι φίλοι της γης, Friends of the Earth και ούτω καθεξής. Τέτοιες οργανώσεις. Εδώ θέλαμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση ευρύτερη ούτως ή άλλως με τους Ευρωπαίους νομοθέτες και γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε ορισμένα κύρια σημεία που μας αφορούν, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στον ιστοτοπό μας κάποιες ιδέες για το ρόλο και την πείρα μας που μπορεί να είναι προφανή ίσως για μια περιβαλλοντική οργάνωση που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Είμαστε συνδεόμενο μέλος της ΣΕΝ και συνεργαζόμενοι με τη ΣΕΝΕΛΕΚ αλλά όχι μέλη στην έτσι. Είμαστε, ε, συνεργαζόμαστε, παρέχουμε μάλλον εμπειρογνώμονες και συνεργαζόμαστε με 40 τεχνικούς φορείς και επίσης παρέχουμε τεχνικές περιβαλλοντικές εμπειρογνωμοσύνες προκειμένου να, να δώσουμε ένα αντίβαρο στην βιομηχανική συμμετοχή σε αυτούς τους φορείς. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τη αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε μέλος του Panel Express και εκπροσωπούμε ένα μέρος της κοινωνίας των πολιτών και του δημόσιου ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Πραγματικά είμαστε μέρος της διαδικασίας τυποποίησης από τα πιο χαμηλά επίπεδα όπως ε, επεσήμανε και ένας συνάδελφος. Και είμαστε και η μόνη περιβαλλοντική οργάνωση που συμμετέχουμε στην όλη προσπάθεια τυποποίησης. Ο στόχος μου είναι να μιλήσω για την επιτάχυνση και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας στη διαδικασία τυποποίησης. Η ΣΕΝ έχει αναπτύξει κάποια χρήσιμα εργαλεία και ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πλαίσιο για να επιτρέψει τη χρήση τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει και κάποια βήματα, σταδιακά βήματα στη διαδικασία, υποχρεωτικά ώστε να διασφαλίζονται κάποιες ε, περιβαλλοντικές μέρημνες το θέμα είναι δηλαδή αν έχουν ληφθεί υπόψη και αν πρόκειται να ληφθούν υπόψη. Η δική μας οργάνωση, η ΕΚΟΣ, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το σχεδιασμό των ε, διατηθέμενων εργαλείων. Βάσει προτάσεων της ΕΚΟΣ, η έκθεση των ε, ειδικών προβλέπει και την σταδιακή χρήση των εργαλείων αυτών, καθώς και το mainstreaming της συμπερίληψης των περιβαλλοντικών μεριμνών στην διαδικασία τυποποίησης. Δηλαδή κάθε προϊόν μπορεί να έχει πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Η συνδυασμό τυποποίηση και τη υλοποίηση των ε, περιβαλλοντικών μα πολιτικών τώρα είναι ζωτική σημασία νομίζω να γίνει σε αυτή τη διάκριση μεταξύ νομοθεσία και τυποποίηση των σχετικών ε, οδηγιών και του πώ ε, θα οριστεί η εντολή για την ανάλογη Επιτροπή Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Αυτό είναι ρόλο που πρέπει να αναλάβει ο Ευρωπαίο νομοθέτης. Κάτι που στο παρελθόν σίγουρα δεν είχε γίνει πάντοτε με επιτυχία. Θα πρέπει λοιπόν τα ανάλογα εργαλεία να χρησιμοποιούνται όταν ε, είναι ρυθμιστική ανάγκη αυτό και θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος των αποτελεσμάτων από τις δημόσιες αρχές, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για τα διάφορα πρότυπα, τα υποχρεωτικά. Η Επιτροπή επίσης θα πρέπει να ελέγχει τις πολιτικές με σοβαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η γεωργία και το καθεξής. Θα Μπορούσα να πω πολύ περισσότερα για τα περιβαλλοντικά, αλλά κυρίως θα ήθελα να μιλήσω για την ε, ενίσχυση και την ε, μεγαλύτερη συμπερίληψη των ε, δημόσιων πολιτικών στην όλη δικασία της τυποποίησης, γιατί αυτό θα ενισχύσει και την περιβαλλοντική, περιβαλλοντική διάσταση. Νομίζουμε ότι η υλοποίηση και η περισσότερη διευκρίνηση της διαδικασία τυποποίηση από του φορεί, του υπεύθυνου φορού, θα πρέπει να περνάει και από τον ανάλογο έλεγχο, του φορεί ελέγχου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον υπάρχουν ε, ενδιαφέροντα διαφορετικά και από το δημόσιο, γιατί οι ιδιωτικοί φορεί ε, κυρίω κινούνται από το οικονομικό συμφέρον. Θα πρέπει λοιπόν το δημόσιο συμφέρον να είναι ο πρώτος, η πρώτη προτεραιότητα της διαδικασίας τυποποίησης. Η εθνικές αρχές ε, κόρησης δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για όλους τους φορείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει με γραπτές συμφωνίες με τη εν και σε τις προϋποθέσεις για την εκχώρηση κάποιων αποφάσεων. Θα πρέπει λόγω χάρη η δημόσια στήριξη να είναι υποχρεωτική για τους εκπροσώπους με δημόσιο, που εκπροσωπούν δημόσια συμφέροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε όλες τις διαδικασίες λοιπόν τυποποίησης θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναφέρθηκε το παράδειγμα των καταναλωτών ε, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι ακόμη πιο χαμηλή η εκπροσώπησή μας σε σχέση με τους καταναλωτές. Εκπροσωπούμεθα μόνο σε ένα κάτω μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΚ Επίσης, έχουμε χρηματοδότηση 25.000 ευρώ από την Επιτροπή των Κατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΟΧ. Αλλά είμαστε χαμηλότερα χρηματοδοτούμενη οργάνωση που παρίσταται σήμερα στην ακρόαση. Τώρα κάποιες βασικές προτάσεις που θα πρέπει να επιτελεστεί περαιτέρω πρόοδος πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι νομοθέτες θα πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά την παραγωγή προτύπων ε, με στόχο της δημόσιας πολιτικές, όπως και ο Στίβεν, ε, σας ε, παραπέμπω και εγώ στο ανάλογο παράρτημα. Θα πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσο υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση στα τεχνικούς φορείς και το συζητήσαμε αυτό και στο επίπεδο και σε ΕΝΕΛΕ και το συζητούμε ακόμα και στους τέσσερις οργανισμούς εκπροσώπησης των Ευρωπαίων εταίρων θα πρέπει να δοθεί μία ψήφο στον καθένα τουλάχιστον για πρότυπα ιδίω τα οποία συνεισφέραμε ενεργά. Επίση, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν δημόσιε συζητήσει για την ελεύθερη διάθεση κάποιων ορισμένων επιμένων βασικών προτύπων και βεβαίω από την άλλη για το ενδεχόμενο αντισταθμίση του απώλεια εισοδήματο για τους φορεί τυποποίηση. Και τέλο, κάτι εξίσου σοβαρό. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα έρθουν οι φραγμοί για πολλέ ε, περιπτώσει πρόσβαση, όπω τα τέλη για τη συμμετοχή σε επιτροπέ και εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων. Θα πρέπει λοιπόν ε, όλοι να μπορούν να εκπροσωπηθούν με τον ίδιο τρόπο εδώ. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και τη δυνατότητα συμμετοχή στην ακρόαση και να κλείσω λέγοντα ότι η κοινωνία των ενδιαφερομένων των πολιτών και των ε, αρμόδιων φορέων θα πρέπει να λάβει την ανάλογη συμμετοχή στην όλη αυτή τη δικασία τυποποίηση. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι συστάσεις σας και τέλος ο κύριος Μπόι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία εκ μέρους του ΕΤΟΥΙ να λάβω το λόγο ενώπιον σα, Είναι πολύ ενδιαφέρον που μπορούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να παρακάθουμε εδώ μαζί με τόσο εξέχοντες συναδέλφους. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για, τα, για τις Εργασιακές ΕΤΟΥΙ, έχει εμπλακεί στην δημιουργία προτύπων σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, και οικονομικά πρότυπα και αυτό μας δίνει μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τους κατασκευαστές και τους σχεδιαστές για το πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε προϊόντα τα οποία είναι πιο ασφαλή από τα γενοφάσκια τους και τα οποία να είναι πράγματι σύμμορφα με τις προσδοκίες των χρηστών. Δεύτερον, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να καλύψουμε το χάσμα το οποίο μας χωρίζει μεταξύ της ε, σχεδίασης και του τόπου εργασίας και να επικυρώσουμε σε επίπεδο τόπου εργασίας τις επιλογές που γίνονται από τους σχεδιαστές. Τρίτο σημείο. Θέλουμε να εργαστούμε στην προτυποποίηση γιατί μαζί με τους κατασκευαστές μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα παραγόμενα προϊόντα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Επομένως, η ασφάλεια στον τόπο εργασίας είναι ένας από τους πυλώνες της κοινωνικής οργάνωσης της αγοράς. Αν θέλουμε λοιπόν να το εξασφαλίσουμε αυτό, πρέπει να έχουμε δύο προϋποθέσεις οι οποίες θα πληρούνται. Μία αξιολόγηση του αντικτύπου και την πλήρη συμμετοχή των εμπλεκομένων. Η καταμέτρηση λοιπόν του αντικτύπου της προτυποποίησης. Εδώ θέλω να ξεκινήσω από την διαφάνεια αυτή, όπου αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την τυποποίηση σε μια σειρά στρατηγικών τομέων όπου μπορεί η τυποποίηση να υποστηρίξει την νομοθεσία. Εδώ βλέπετε και μία επιλογή τομέων. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η ασφάλεια και η υγεία στον τόπο εκατομμύριων εργαζομένων <clears throat> καλύπτεται από ένα συνδυασμό οδηγιών για εναρμόνιση προϊόντων και επίσης οριζόντιων οδηγιών για τα κοινωνικά θέματα. Περνάμε στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε λοιπόν από τη μία μεριά νομοθετικές ρυθμίσεις για κοινωνικά θέματα αλλά και οδηγίες για τα, για τα ίδια τα προϊόντα. Αυτό ο συνδυασμό πιστεύω ότι λειτουργεί πολύ καλά για να εξασφαλίσει υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασία και πιστεύω ότι αν η τυποποίηση εμπλακεί στα θέματα αυτά και αν έχει σαν στόχο να υποστηρίξει την νομοθεσία, τότε η τυποποίηση δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει αρνητικά στο τωρινό κανονιστικό πλαίσιο για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασία. Γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγάλη σημασία στη διαδραστική επιφάνεια μεταξύ της τυποποίησης και των ρυθμίσεων στον τόπο αυτό της αγοράς. Ένας δεύτερος πυλών η συμμετοχή των εμπλεκομένων. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ότι δεν υπάρχει έναυσμα για τους ε, χρήστες το οποίο να είναι συγκρίσιμο με το οικονομικό συμφέρον των κατασκευαστών και της βιομηχανίας που οι τελευταίοι καθορίζουν τη διαδικασία και είναι θεμητό ότι αυτοί θα πρέπει να κατευθύνουν τη διαδικασία, αλλά για τους καταναλωτές, για τους ε, ε για το περιβάλλον, για τα εργατικά συνδικάτα, δεν υπάρχει άμεσο μέρισμα σε οικονομικό επίπεδο από αυτή τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η έλλειψη ισορροπίας έχει σαν αποτέλεσμα ότι δεν βρίσκονται όλοι με την ίδια δύναμη διαπραγμάτευσης στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, το συμπέρασμα είναι ότι τα πρότυπα τα οποία προκύπτουν μπορεί να μην έχουν αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα και να μην ενσωματών τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πιο ασθενών εμπλεκομένων. Τώρα, δεν πρέπει να μας εκπλήσει η ύπαρξη αυτής της έλλειψης ισορροπίας, αλλά αυτή είναι μια εγγενής έλλειψη ισορροπίας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας, σε ό,τι αφορά την διαπραγματευτική ικανότητα, αυτή πρέπει να επιληθεί με κατάλληλα μέτρα, ιδίω όταν τα πρότυπα υποστηρίζουν την νομοθετική διαδικασία. Προσκαλούμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να κατανοήσει ότι οι κυβερνήσει θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για να θεσπίσουν προποθέσει για τυποποίηση η οποία πράγματι αντανακλά τι ανάγκε τη κοινωνία. Μπορούμε να επιτύχουμε λιγότερη ρύθμιση μέσα από την προτυποποίηση. Εμείς θα υποστηρίξουμε πάντα την προτυποποίηση σε τομείς που ενδιαφέρουν το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία με την προϋπόθεση ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν την απαραίτητη δομική υποστήριξη στο κατάλληλο επίπεδο. Όταν όμως περνάμε από τις τεχνικές και στις λιγότερο τεχνικές ε, προτυποποιήσεις έχουμε άλλες προκλήσεις. Γιατί τίθεται εδώ και το θέμα πρώτον της εγγενού ασφάλειας ότι πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνεται το θέμα της ασφάλειας σε όλα τα προϊόντα. Αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί μία ε, συνένεση ακόμα και σε σχέση με την σχεδίαση των προϊόντων, την μηχανολογία των προϊόντων. Και φυσικά όταν περνάμε από διατάξεις για υλικά αγαθά σε άειλα αγαθά, είναι πολύ δύσκολο να, δούμε, να, να βρούμε μία συνένεση. Δεύτερον, για τα προϊόντα. Η εποπτεία της αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε ποια προϊόντα είναι ελληματικά και έχουν προβλήματα ασφάλειας. Όταν όμως είμαστε στον τομέα το μη βιομηχανικό, αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο εργαλείο για να δούμε τα λανθασμένα πρότυπα. Τέλος. Μόνο με μία ισορροπημένη παρουσία των εμπλεκομένων μπορεί η τυποποίηση πράγματι να μας οδηγήσει σε καινοτομίες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία να λάβω το λόγο ενώπιόν σας και είμαι έτοιμος να απαντήσω οποιαδήποτε ερωτήματα μου απευθυνθούν. Well, thank you very much ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπόη και εμείς χαρήκαμε που σας ακούσαμε για το τελευταίο που είπατε, να σας διαβεβαιώσω πως η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την υποπτία της ε, αγοράς με βάση τα όσα είχε κάνει στο παρελθόν η κυρία Σχάλντε Μόζε και οπότε δεν ε, είναι βεβαίως θέμα της σημερινής αλλά παρόλα αυτά το σύστημα που ε, θα δημιουργήσει ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα για τους καταναλωτές είναι κάτι που μας απασχολεί, οπότε η συνεισφορά σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους συναδέλφους. Ο εισηγητής, ο καθηγητής ο κ. Δεκάμπος επίσης και η κυρία Κόμη και η κυρία Ρούλε. Λοιπόν, σύντομα, οπότε να τελειώσει ο πέρα κατάλογος των ομιλητών. Λοιπόν, Κόσιτσικ. Σύντομη ερώτηση προς τον ε, Ραλφ Λότες. Αναφέρατε στην παρουσίασή σας πως ε, πρέπει να υπάρχουν κάποια ε, κάποιες βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να είναι δωρεάν για το κοινό. Μπορείτε να μου πείτε ποιες εννοείτε. ένα λεπτό έτσι ενδεικτικά συνάδελφοι, ο καθηγητής ε, κύριος Ντεκάμπος. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές ε, για τις ε, συνεισφορές τους σε αυτή την συζήτηση. Θα ήθελα να απευθύνω ερώτημα προς τον Στέφαν Μπόι για τα ζητήματα της ασφάλειας στην εργασία. Όλοι βεβαίως συμφωνούμε με την σημασία της ε, συμμετοχής σε κάθε φάση της κατάρτισης των προδιαγραφών, ε, συμμετοχής των εργαζομένων. Το ερώτημα είναι πως σε πολλές χώρες υπάρχει μείωση του ενδιαφέροντος των συνδικάτων και θα ήθελα να πει ο Στέφανο εάν ε, κάτι τέτοιο ισχύει. Η αίσθησή μου είναι πως αυτό είναι γιατί περνάμε από μια κοινωνία βιομηχανική σε μια κοινωνία υπηρεσιών και αυτό έχει σαφείς ε, συνέπειες. Οπότε η τυποποίηση των υπηρεσιών όπως ε, παραδείγματο χάρη η εκπαίδευση, η κίνδυνη στην εκπαίδευση, η βία στα σχολεία και στα νοσοκομεία είναι κάτι που είναι δύσκολο να τυποποιηθεί δηλαδή ποιο είναι το επίπεδο του κινδύνου και των μέτρων, αλλά είναι κάτι το δυνατόν. Το ερώτημα μου είναι, συμφωνείτε με αυτή τη μείωση που βλέπω εγώ. Θεωρείτε, αν συμφωνείτε, πώς θεωρείτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διμερείς ευθύνες και των επιχειρηματιών και των υπολείπων εμπλεκομένων. Ευχαριστώ όλα ακόμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο ερώτημά μου. Δηλαδή η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και η βελτίωση του νομικού πλαισίου. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή των τελικών χρηστών για τα θέματα αυτά. Η έκθεση που αναφέρθηκε τόνισε ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι η εξέλιξη των ε, προτύπων θα μπορούσε να γίνει μονάχα επί τη βάση του πραγματικού ωφέλους το οποίο θα πρέπει να καταδειχθεί. Και φυσικά, όπως είπε και ο κύριος Ράσελ, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν και οι καταναλωτές στην ανάπτυξη συστημάτων τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο στόχος μας λοιπόν θα πρέπει να είναι τα συστήματα αυτά να εκπροσωπήσουν απόλυτα και το συμφέρον και την άποψη των καταναλωτών και των τελικών χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της δημόσιας ε, της έλλειψης δημόσιας παρουσίας, της ε, ιδιωτικής λοιπόν λειτουργίας, παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επομένως, για μας είναι απαραίτητο να υπάρξει η προστασία και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν... Δεν το βρίσκω τέλο πάντων. Ρώτησα και πριν για τη συμμετοχή των ε, διαφόρων οργανώσεων στον εθνικό τομέα και η απάντηση ήταν πως ε, θα πρέπει να γίνει αυτό μέσω της συμμετοχής ε, από το ίντερνετ. Έχετε σχετικές εμπειρίες και ποιες ήταν αυτές και αν είναι μια δυνατότητα αυτή για την βελτίωση της συμπερίληψης οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων κτλ. Το ένα ερώτημα ήταν αυτό. Το άλλο ερώτημα είναι το θέμα της διαφάνειας. Λέτε πως όταν έχουμε υποχρεω... υποχρεώσεις πρέπει να τα επιτηρεί αυτά ο νομοθέτης, αλλά υπάρχει η σχετική οδηγία που λέει πως ε, θα πρέπει ε, να μαθαίνουμε όσο δυνατόν λιγότερες πληροφορίε για τις πρωτεγραφέ. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η διαφάνεια. Και τέλος ε, υπάρχουν παράπονα για τη μεγάλη διάρκεια αυτή της διαδικασίας. Ξέρετε πώς μπορεί να μειωθεί αυτή η διάρκεια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ ως πρόεδρος να θέσω ένα ερώτημα προς όλους με βάση αυτό το οποίο είπε ο Στίβεν Ράσελ για την πρότασή του για αυτό το οποίο σε μια εναλλακτική γραμμή παραγωγής για προδιαγραφές με δημόσιο συμφέρον. με αν το υποστηρίζουν όλοι αυτό και από αυτό το οποίο Στίβεν για το πώς θεωρεί ότι μπορεί κάτι τέτοιο να ενταχθεί στις προτάσεις που υπάρχουν επιτάπητος. Λοιπόν, θα ζητήσω τώρα τους τρεις ομιλητές μας να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, βρήκαμε λίγα χρόνο, αλλά ούτως ή άλλως θα υπάρχει το ρολόι. Ε, οπότε δύο λεπτά παρακαλώ ο καθένας. Στίβεν Ράσελ λοιπόν παρακαλώ πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω ε, τις απαντήσεις. Πρέπει να τονίσουμε πως ε, εμείς στην ΑΝΕΚ υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή τυποποίηση πλήρως, όπως ανέφερα μας έχει βοηθήσει στο να δημιουργήσουμε την κοινή αγορά και η κοινή αγορά έχει ωφέλη για τις καταναλωτές. Αυτό είναι αναμφίβολο. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στην ιδιωτικοποίηση της νομοθεσίας, όπως λέγεται, είναι μία διασφάλιση πως το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται στην διαδικασία αυτή. Θα ήθελα να τονίσω πως εμείς θεωρούμε πως συμπληρώνουμε την βιομηχανία σπάνια ε, συγκρόμαστε μαζί της. Όσον αφορά την εμπλοκή μέσω διαδικτύου, Βεβαίω το σύστημα γίνεται πιο διαφανές και το ζήτημα είναι βεβαίω η εμπειρία. Εάν δεν υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις με εμπειρία δεν έχει νόημα να μιλάμε και για συμμετοχή από το ίντερνετ. Είναι σαν να έχουμε ε, εκπροσώπηση ατόμων. Πρέπει να είναι οι άνθρωποι ειδικοί για το χρόνο που χρειάζονται οι διαδικασίες ε, στο παρελθόν, στην ΣΕΝ, ήμουν υπεύθυνο για το τριετέ πλαίσιο ανάπτυξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Μπορεί να σα ακούγεται πολύ αυτό, αλλά παλαιότερα οι προδιαγραφέ χρειάζονταν 7 έω 8 χρόνια κατά μέσο όρο. Οπότε και τα τρία χρόνια ακούγονται μεγάλο διάστημα, αλλά λάβετε υπόψη το πόσο χρειάζεται να δημιουργηθεί η νομοθεσία. Γι' αυτό και το 1985 εισήχθη η νέα αυτή προσέγγιση γιατί η Κομισιόν και τα θεσμικά όργανα δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν την ε, ενιαία αγορά με την νομοθεσία και στράφηκαν στις προδιαγραφές. Αν μου δώσετε άλλα 30 δευτερόλεπτα για την ε, γραμμή αυτή παραγωγή στην δεύτερη πρέπει να γίνει εντός του συστήματος, δεν πρέπει να αλλάξει το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης που υπάρχει πρέπει να αναπτυχθεί όχι από εθνικές αντιπροσωπείες αλλά από ε, ενδιαφερόμενους, αλλά ούτως ή άλλως οι, εθνικές, ε, εθνικοί φορείς θα ψηφίζουν και θα τα δημοσιεύουν ως εθνικές πρωτεγραφές. Αυτή είναι λοιπόν, αυτός είναι ο εθνικός έλεγχος. Και θεωρούν πως η Επιτροπή 9834 που ήδη κρίνει τις εντολές για τους φορείς ε, τυποποιήσεων θα μας πει εάν θα ακολουθήσουμε τον εθνικό δρόμο ή τον δρόμο της συμμετοχής των Σα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που το διευκρινίζετε αυτό. Ο κύριος Λότες. Εύρη, θα ήθελα καταρχήν να υποστηρίξω όλα αυτά τα οποία είπε ο Στίβεν και θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο στο θέμα που έθελε ο κύριος Κούσνετσεκ σε μένα. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα για την ευκαιρία πρέπει να είναι κανείς σύντομος και να δώσει τα κύρια σημεία σε μια τόσο σύντομη παρουσίαση. Η ελεύθερη ε, διάθεση των προτύπων είναι ένα από τα πιο επίμαχα θέματα από το πάνελ. Κανείς δεν έχει βρει μια κατάλληλη λύση. Τα αποτελέσματα, οι συνέπειες είναι σαφείς για το σύστημα. Όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για αυτό το θέμα. Αλλά και από άποψη διακυβέρνηση της διαδικασίας προτύπων είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς στους πολίτες ότι πρέπει να πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση σε κείμενα τα οποία είναι σημαντικά πρότυπα, είναι σημαντικά για την συμμόρφωση με την νομοθεσία. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν να ξέρουν οι πολίτες με ποιες διαδικασίες εφαρμόζεται αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα διακυβέρνησης ποια είναι τα κύρια πρότυπα, τα κεντρικά πρότυπα. Αυτό πρέπει να το φασίσει ο νομοθέτης και θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει με μερικά τα οποία τα έχει εντοπίσει η ίδια η νομοθεσία και να δούμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες της αλλαγής της διαδικασίας. Αν μπορώ να κάνω μια πρόταση όμως, ένα πάρα πολύ επίμαχο θέμα σε διεθνές επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι το θέμα του καθορισμού των νανοθέσεων που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας, ένα στάνταρ της ISO. Σε ποιο σημείο λοιπόν θα παρέμβει η νομοθεσία για την νανοτεχνολογία ή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την νομοθεσία του REACH που καλύπτει τις χημικές ουσίες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό για τους πολίτες να ξέρουν <clears throat> πώς θα λειτουργήσει και πώς θα διατυπωθεί ο ορισμός για τις νανοθέσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας προτύπων που θα πρέπει να τύχουν απόλυτα δωρεάν διάθεσης προς το κοινό. Ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος Μπόιντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι έκαναν κάποια πολύ ενδιαφέροντα ερώτηματα. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σαφής. Η εργασιακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτεται από νομοθεσία με ελάχιστε απαιτήσει. Κάθε κράτο μέλο βασίζεται στην παράδοσή του, την οικονομία, του ε, κανόνε που επικρατούν και τι πόρου του. Μπορεί να κάνει περισσότερα από τι ελάχιστε απαιτήσει, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε κράτο μέλου. Όμω σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει και το συμβουλευτικό σώμα. Ένα τριμερή οργανισμό που ασχολείται με, τον, ε, με την εργασιακή ασφάλεια και υγεία σε οριζόντιο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για την ε, μείωση του ενδιαφέροντο των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην ε, εργασιακή ασφάλεια και υγεία. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, διότι δεν έχουμε καταμετρήσει ακόμη την αλλαγή από τη βελτίωση των συνδικών ασφάλεια και υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει των στατιστικών, Έχουμε ακόμη 6.000 ε, ατυχήματα θανάσιμα ετησίω στο στον εργασιακό χώρο. Επίσης έχουμε προβλήματα με τις, μυο... με τις μυϊκές ε, παθήσεις και αυτό ε, δείχνει και το πώς αλλάζουν τα πράγματα από το πέρασμα σε μια από τη βιομηχανική στην ε, οικονομία των υπηρεσιών. Εάν οι διμερείς συμφωνίες για τον εργασιακό χώρο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων παραμείνουν ως έχουν, τα εργαλεία τυποποίησης μπορούν να φέρουν τη διαφορά προκειμένου να έχουμε οριζόντια συγκρίσιμα μεθοδολογικά εργαλεία για να αποτιμούμε τον κίνδυνο. Αυτό θα είναι όμως ένα ξεχωριστό έργο. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι από κοινού θα, δουν, θα εντοπίσουν τα ωφέλη. ακόμη και σε ένα πλαίσιο που η αγορά ασκεί πιέσει, όπου υπάρχει πίεση στην αγορά απασχόληση, που υπάρχει πίεση για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και περισσότερα προϊόντα, που χρειάζεται η ανάλυση κόστου ωφελία. Και παρόλο που έχουμε να κάνουμε με οικονομικού όρου, και κοινωνική στόχη πρέπει να είναι συμβατή και σε εθνικό επίπεδο και πρέπει αυτό να γίνει και σε ευρωπαϊκό. Η τυποποίηση μπορεί πολλά να προσφέρει ως προς τα συγκρίσιμα εργαλεία μεθοδολογίας για να βελτιώσουμε τη στατική μας. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. I think... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για αυτά τα οποία μας είπατε. Νομίζω πως όλοι αξίζεται άλλο ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Uh, θα περάσω τώρα στο τελευταίο κομμάτι και μετά θα έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις υπό το γενικό θέμα η στρατηγική σημασία της τυποποίησης για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα ακούσουμε κάποιους ειδικού που είναι βεβαίως ε, σε κάποιους οργανισμούς που εφαρμόζουν ε, αυτές τις πρωτεγραφές. Έχουμε λοιπόν τον Έντρια Χάρης, Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Βιομηχανιών ε, με μηχανικής. Επίσης τον Λουκά Γκουρτζογιάννη του με του Ευρωπαϊκού Γραφείου Μικρομισών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, την Μπεθ Στάμφλ Μπλάχα που θα μιλήσει για τις υπηρεσίες και που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, τον Μάρκους Ράιγκλ, πρόεδρο της ομάδας εργασίας ε, τυποποίησης για το Γερμανικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών και τον Γιώχεν Φρίντιχ που ήταν εκπρόσωπος στην ε, Επιτροπή για την τεχνολογία επικοινωνιών και πληροφορικής. Και πάλι λοιπόν έχετε 7 λεπτά. Ελπίζω να μπορέσετε να τηρήσετε και εσείς το χρόνο όπως οι προηγούμενοι. Θα δώσω τώρα τον λόγο πρώτα απ' όλα στον Adrian Χάρης. Καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Τσόσνικ για την σημερινή ε, πρόσκληση και είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία η συνεδρίαση αυτή γιατί και η Κομισιόν ετοιμάζει βεβαίως σχετική νομοθεσία, αλλά και δεν παίζει και αγώνα στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ποιοι είμαστε. Είμαστε ένα σύνδεσμος με μέλη από 22 χώρε. καλύπτουμε γύρω στο 28% τη βιομηχανική παραγωγής της Ένωσης και μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών. Ένα σημαντικός ε, τομέας, ε, απασχολεί πολλού ανθρώπου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τυποποίηση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι πως από τη δική μας την Σκοπιά θεωρούμε πως είμαστε εμπλεκόμενος και είμαστε ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της τυποποίησης μακράν και από πλευρά συμμετοχή και από πλευρά χρημάτων και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε επόμενη διαφάνεια. Οπότε προφανώς αν έχουμε τέτοια ανάμειξη είναι γιατί υπάρχουν σαφή ωφέλη για τη βιομηχανία, επιταχύνει το άνοιγμα νέων αγορών, ας δούμε παραδείγματος χάρη τι γίνεται τώρα με τα ηλεκτρικά οχήματα, μια νέα αγορά που πιθανώς θα αναπτυχθεί και η τυποποίηση θα παίξει ρόλο κλειδί και ελπίζω το απόγευμα μάλλον όχι την ερχόμενη εβδομάδα νομίζω θα έχουμε την εντολή τυποποίησης για τα ηλεκτρικά οχήματα από την Κομισιόν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για εμάς για να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων αγορών, γιατί αυτή είναι βεβαίως η βασιλική οδός. Επίσης ευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά, π.χ. έχουμε τέσσερα άτομα στην Κίνα που φροντίζουν ε, ακριβώς ε, στην προώθηση διεθνών προδιαγραφών και καλωσορίζουμε τη στήριξη της Κομισιόν που έχει και γραφείο στην Κίνα με ειδικού ε, στην τυποποίηση και προσεχώς και στην Ινδία. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ γιατί η τυποποίηση παίζει ένα ρόλο κλειδί σε εμπορικέ μα δραστηριότητε. Ε, έχει λέει, μεγάλη σημασία για την αγορά επίσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαφές νομίζω αυτό για τις μικρές εταιρείε. Ε, δίνει πρόσβαση στην γνώση, στην πιο τελευταία γνώση και βοηθάει τις εταιρείες που συμμετέχουν να είναι πιο ανταγωνιστικές. Βεβαίως, όλοι μιλάνε για την εκπροσώπηση των συμμετεχόντων και σαφώς υπάρχουν ωφέλη ε, για τους καταναλωτές στην τυποποίηση. Το πρώτο που αναφέρθηκε είναι η διαλειτουργικότητα, δεύτερον βεβαίως είναι η εμπιστοσύνη και τρίτον είναι το κόστος. Πρέπει να θυμόμαστε πως ε, το κόστος μειώνεται λόγω της εσωτερικής αγοράς, οπότε η τυποποίηση είναι πρώτα απ' όλα ένα εργαλείο που επινοήθηκε από τη μηχανία πριν από πολύ καιρό για να έχει πρόσβαση στις αγορές και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Θα δώσω κάποια παραδείγματα κανονισμών. Ο βασικός κανονισμός ε, βεβαίως ε, ορίζεται ε, από τους πολιτικούς όπως θα έπρεπε και εφαρμογές στα προϊόντα από την τυποποίηση. Και πάμε και πέρα από το προϊόν γιατί έχουμε και την επιτήρηση της αγοράς που ζητάει προδιαγραφές και αυτό έχουμε κάνει και ελπίζουμε να συνεχιστεί η συνεργασία. Τώρα, επόμενη διαφάνεια, κάτι το οποίο είναι σαφές νομίζω και πρέπει να γίνει ξεκάθαρα, είναι πως οι προδιαγραφές δεν είναι νόμοι, γιατί υπάρχει σύγχυση συχνά στο μυαλό των ανθρώπων που ταυτίζουν τα δύο. Οι δεν είναι ε, δεν αναπτύσσονται ε, για αυτό το στόχο, πρώτο και κύριο λόγο έχουν την αγορά. Οπότε αναπτύσσονται από τους χρήστες, δηλαδή τις εταιρείε για τον σχεδιασμό των προϊόντων, τις δοκιμές, τις μετρήσεις κτλ. Σε ένα χαμηλότερο επίπεδο βεβαίω βλέπουμε πως οι προδιαγραφές είναι εθελοντικές όσον αφορά και την συμμόρφωση και υπάρχει ένας απλός τρόπος για να θεωρούν πως κάποιος συμμορφώνεται. Αυτό είναι θετικό γιατί έχουμε ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα νομικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως η Κομισιόν μιλάει για απλοποίηση, αλλά αν δείτε την νομοθεσία που αφορά τα προϊόντα δεν είναι καθόλου απλή. Οπότε χρησιμοποιούνται ως ένα εργαλείο αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ε, αλλά δεν θέλουμε να γίνει κάτι το υποχρεωτικό, γιατί το να χρησιμοποιηθεί ως ένα τέτοιο εργαλείο όπως ε, κάνουμε για προϊόντα μεγάλης ε, κλίμακας ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά όταν έχουμε ένα με μόνο με ένα προϊόν ή σχέδιο μηχανικό, κάτσο που είμαστε πρωταθλητές οι Ευρωπαίοι, μπορεί ο καθένα να κάνει το δικό του σχέδιο, τι δικέ του προδιαγραφέ και το δικό του τεχνικό φάκελο για να δικαιολογήσει γιατί επέλεξε κάτι το συγκεκριμένο. Συμπερασματικά λοιπόν για εμάς το Ευρωπαϊκό Σύστημα χρειάζεται δημόσια στήριξη και όχι γραφειοκρατικό έλεγχο. Η ζωτικότητά του είναι κάτι που εξαρτάται από μια κάποια ελευθερία. Στον τομέα της νομοθεσίας προϊόντων και υπηρεσιών θα θέλαμε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των κοινωνικών απαιτήσεων που βεβαίως θα τις κρίνουν αυτοί που καθορίζουν την πολιτική οι ρυθμιστικές αρχές το τι θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθήσει η κοινωνία, είτε μιλάμε για υγιεινή και ασφάλεια, περιβάλλον, ενέργεια και επαφίεται μετά στο σύστημα τυποποίησης να κάνει αυτή την υποστηρικτική λειτουργία όσον αφορά την ανάπτυξη των προϊόντων, τις δοκιμές ε, και τις μετρήσεις. Δεν πρέπει να ανακατεύσουμε αυτά τα δύο. Από τη δική μας σκοπιά, αν θέλουμε να ενισχύσουμε το σύστημα τυποποίησης, αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από τους ενδιαφερόμενους ε, και αυτό σημαίνει πως η ανάπτυξη πρέπει να γίνει στο εθνικό επίπεδο. Όσο ελκυστικές και αν είναι οι Βρυξέλλες, είναι απλούστερο για τις περισσότερες εταιρείες να εργάζονται σε τοπικό επίπεδο, στη δική τους γλώσσα, να συμμετέχουν. Λοιπόν, εκεί είναι λογικότερο, γι' αυτό εκεί πρέπει να εστιάσουμε και ελπίζω να συνεχίσει να υπάρχει στήριξη στην ανάπτυξη σε αυτό το επίπεδο και να αυξηθεί η εκπαίδευση και η ενημέρωση στο, στην γλώσσα του καθενός και στους ανθρώπων που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις προδιαγραφές. Ευχαριστώ. The next time, very Κατόπιν ε, χαίρομαι που ορίζω τον Λουκά Γκουρτσογιάννη, εξ ονόματος της Νορμάπμε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά για την ευκαιρία αυτή που μα δίνεται να συζητήσουμε τα ζητήματα προτυποποίηση που είναι πολύ σημαντικά για μα. Ακολουθώ τον κύριο Χάρη και μπορώ να τονίσω ότι είναι οι τέσσερι είναι κύριοι τομεί στου οποίου εργαζόμαστε. Η προτυποποίηση είναι πολύ σημαντική λοιπόν σε αυτού του τομεί και απλώς θέλω, εν συντομία, να σας δείξω τι κάνει η Νορμάπμε. Είναι ένας φορέας μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τονίζω μόνο μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπροσωπεί τομεακή και εθνική συμμετοχή. Περίπου 4 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκπροσωπούνται και με, μέσω μιας συμβάσεως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς εκπροσωπούμε και τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για καθαρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτή είναι η πιο αδύναμη εμπλεκόμενη. Γι' αυτό υπάρχει υποστήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην επόμενη διαφάνεια δείχνω ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα τυποποίησης έχουν ήδη καταγραφεί και τεκμηριωθεί από προηγούμενες μελέτες που δεν χρειάζεται εδώ να επεκταθώ ιδιαίτερα. Η έλλειψη οικονομικών και ανθρωπινών πόρων για μικρές εταιρείε δεκατών. Φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι εμπειρογνώμος στα θέματα τυποποίησης. Η δυσκολία να βρεθούν και να υπάρχει πρόσβαση στα πρότυπα. Θέλω να πω και κάτι για τη δυσκολία κατανόησης των προτύπων. Τα πρότυπα πολλές φορές γράφονται σε μια ιδιαίτερα πολύπλοκη γλώσσα και φρασιολογία. Ακόμα και όταν μεταφραστούν στην μητρική του γλώσσα του καθενός, πάλι δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ιδιαίτερα τις ε, διατυπώσεις, τα διπλά ολοκληρώματα, τις άπειρες σειρές κτλ. Όλα αυτά απαιτούν μια μετάφραση από εμπειρογνώμονες που μπορεί να γίνει σε μεγάλες εταιρείες αλλά όχι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε καν σε φορεί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί και οι φορεί μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν τα ίδια προβλήματα δυσκολιών με υλικού και ανθρώπινους πόρους. Τα πρότυπα εφαρμογή επίση μπορούν να είναι δύσκολα, γιατί χρειάζεται κανείς να επενδύσει σε εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και σε νέα συστήματα παραγωγή. Και τέλος, η συμμετοχή είναι πολύ δύσκολη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. <clears throat> Χαίρομαι που τώρα βλέπουμε τη δυνατότητα συστημάτων διαδικτύου για την ε, παροχή γνωμοδότησης. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει διαδικασία ψηφοφορία σε πολλά επίπεδα για την τυποποίηση. Δεν πρόκειται μονάχα για το να μπορούμε να στέλνουμε την άποψή μας σε ευρωπαϊκά θέματα, αλλά να συμμετέχουμε το σημαντικό είναι και στους φορείς που θα λάβουν την τελική απόφαση. Γι' αυτό λοιπόν παρά τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών είναι ακόμα σημαντική η διαδικασία συμμετοχής. Δυστυχώς η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδηγεί σε διαμάχες. <clears throat> Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή αλλά δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Το γράφημα αυτό προκύπτει από μια ανάλυση 100 τεχνικών περίπου επιτροπών στα πλαίσια της ΕΝ για να δούμε αν χρειαζόταν να παρέμβουμε περισσότερο για την ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα δύο τρίτα των συμμετοχών είναι από εθνικούς φορείς πρότυπων, αλλά εδώ σας δείχνω το 1 τρίτο αυτών που είναι μέλη στους καταλόγους αποστολής email. Δεν είναι οι κατάλογοι συμμετοχής, γιατί αυτούς τους καταλόγους συμμετοχής δεν μπορούμε εύκολα να τους βρούμε στο ίντερνετ και στις ιστοσελίδες. Βλέπουμε εδώ όμως ότι είναι πολύ χαμηλή η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να τονίσω. Προσπαθήσαμε να <clears throat> χωρίσουμε τις διάφορες ε, επαγγελματικές κατηγορίες όπως είναι οι σύμβουλοι και οι επαληθευτές κτλ που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά, γιατί και αυτοί λένε ότι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και αυτοί έχουν κάθε συμφέρον να ενισχύσουν το ρόλο τους με το να προσθέτουν αναγκαιότητες ε, επαλήθευσης ή παροχής συμβουλών. Πρέπει λοιπόν οι λεγόμενες παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποχωριστούν από τη διαδικασία έλεγχου και επαλήθευσης. Σας ανέφερα επίσης ότι στην προσπάθεια του να δούμε τι γίνεται με την προτυποποίηση και τις τεχνικές επιτροπές σε εθνικό επίπεδο για τις 40 ε, περιπτώσεις στις οποίες εμείς έχουμε συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε 12 <clears throat> περιπτώσεις που δεν πήραμε αποφάσεις και 4 αποφα... απαντήσεις που ήταν κάπως φοβεριστικές. Μας είπαν ότι εδώ πρόκειται για θέμα προστασίας της ιδιωτικότητος που δεν μας επιτρέπει οι κατάλογοι των συμμετοχόντων να δημοσιευθούν. Αν υπάρχει σε εθνικό επίπεδο τέτοια νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει την κατάργησή τους, γιατί εδώ μιλάμε για θέματα δημοσίου συμφερόντος. συμφερόντος. Είχαμε μόναχα πέντε χώρες που μας έδωσαν στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα, μας έδωσαν, δείξαν τη χαμηλή συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θέλω να προεκβάλλω τώρα αυτά τα στοιχεία γιατί είναι μονάχα από πέντε χώρε, αλλά αυτά μα δίνουν την εικόνα που σα έδωσα προηγουμένω. Και έρχομαι τώρα στι συστάσει. Πιστεύω ότι μαζί με του άλλου αδύναμου συμμετέχοντες που ανεφέρθηκαν προηγουμένω, είναι απαραίτητο να υπάρξει θεσμική αναγνώριση και υποστήριξη αυτών των ε, συμμεταχόντων στο επόμενο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης Επίσης πρέπει να υπάρξει διατήρηση της χρηματοδότησης και για την ΟΡΜΑΠΜΕ και για τους άλλους ασθενείς συμμετέχοντες. Πιστεύουμε ότι χρειάζονται και δικαιώματα ψήφου και σε επίπεδο BT, TC και σε τελικό επίπεδο. Γιατί δεν μπορεί πάντα να ακουστεί η φωνή των πιο αδύναμων εμπλεκομένων που περνά που να μπορέσει να περάσει από εθνικό επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε δικαιώματα ψήφου σε αυτά τα επίπεδα. Θέλουμε επίση το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίηση να υπάρξει νομική αναγνώριση του δημοσίου συμφέροντος και από την άποψη αυτή οι αρχές του ΠΟΕ, ιδιαίτερα της διαφάνειας και της αμεροληψίας, θα πρέπει να εφαρμοστούν. Για τη διαφάνεια και την αμεροληψία. Εδώ θα πρέπει να συνδεθούν αυτές με την ανάγκη να υπάρξει ένα σύστημα για μη ισορροπημένη ε, συμμετοχή στους φορείς που παίρνουν απόφαση. Επίσης θέλουμε να υπάρχουν ε, εκπτώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επί τη βάση του, του μεγέθους τους για τα πρότυπα, για την πρόσβαση στα πρότυπα που είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος χρειαζόμαστε χρηματοδότηση και υποστήριξη για συμμετοχή, εκπαίδευση και τη χρήση των προτύπων και πάλι σε εθνικό επίπεδο. Και υπάρχουν πολλά πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα θα διατυπώνονται με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι χρήσιμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να είναι δυνατόν να τα κατανοήσουν και έτσι με την εφαρμογή των προτύπων αυτών από τι μικρομεσαίε επιχειρήσει μπορούμε να αυξήσουμε την αναγνωριστικότητα του και την εν γέννη τη ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Well, I was very indulgent. Δεν έδειξε αυστηρότητα ω προ το χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντικέ μικρομεσαίε επιχειρήσει, ω πιο αδύναμο ε, συμμετέχων εδώ στην όλη διαδικασία. Και τώρα με ιδιαίτερη χαρά να δώσω το λόγο στην κυρία Στάμφιλ Μπλάχα, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Αυστριακής ε, Τυποποίησης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί ο Επίτροπος Ταγιάννη είπε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης για τα Προϊόντα είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Θα μπορούσε αυτό όμως που έχει ισχύσει με επιτυχία για τα προϊόντα να μεταφερθεί και στις υπηρεσίες θα μπορούσε κάτι το οποίο είναι μη υλικό όπως οι υπηρεσίε να τυποποιηθεί. Νομίζω αυτά θα μπορούσαμε να τα απαντήσουμε με κάποια πράγματα από την πραγματικότητα αυτά, και στην οθόνη πολλές υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί σε πολλές χώρες και σε διάφορους τομείς βάσει των ετοιμάτων των ε, ενδιαφερομένων και χάρη στην συνεισφορά των ε, ενδιαφερομένων. Έχουμε λοιπόν πρότυπα για, το management και τις συμβουλευτικέ υπηρεσίες, για τα στέγαση, για τον έλεγχο των ε, φυτοφαρμάκων, για τις ναυτικές υπηρεσίες, τις ταχυδρομικές. Όλα αυτά, λόγω της απελευθέρωσης, Επίσης και για τις ε, υπηρεσίες εργολάβων κηδιών. Τυποποίηση λοιπόν των υπηρεσιών. Ναι, μπορεί να γίνει. Το ερώτημα όμως είναι αν θα έπρεπε να τυποποιηθούν οι υπηρεσίες. 70% της συνολική απασχόλησης βασίζεται στις υπηρεσίες της αγοράς και αυτό εκπροσωπεί ένα αυξανόμενο μέρος του ΑΕΠ. Η καινοτομία, η βασική κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης προέρχεται ακριβώς από αυτές τις υπηρεσίες και μέσω των υπηρεσιών. Μιλάμε εδώ για υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με προϊόντα. Αυτό ήδη έχει αναγνωριστεί σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα εγγράφων από το πρόσφατο χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την τυποποίηση και την καινοτομία, που τονίζουν το καινοτόμο δυναμικό που υπάρχει στον τομέα των υπηρεσιών και παραθέτω εδώ την ανάγκη να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα ενδεχόμενα ωφέλη και αυτό σε σχέση με την οδηγία για τι υπηρεσίε. Και κοιτάζοντα προ το μέλλον, η στρατηγική τη Ευρώπη του 2020 υπογραμμίζει, και εδώ παραθέτω, ότι η ανάτηση νέων υπηρεσιών στην υγεία, την ευθύνη μηχανική και ούτω καθεξής δείχνουν ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό για την Ευρώπη και ότι το δυναμικό αυτό θα αξιοποιηθεί μόνον αν αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό. Πού υπάρχει κατακαιρματισμό λοιπόν. Αν δούμε τι παραδοσιακέ υπηρεσίε, θα δείτε ότι υπάρχει διαφορετικό βαθμό ρύθμιση. Όπω για τι μεσαιτικέ υπηρεσίε. Εκεί στα παλιά κράτη-μέλη υπάρχουν κανόνε, αλλά δεν υπάρχει απολύτω τίποτε στα νέα κράτη-μέλη. Η τυποποίηση λοιπόν εδώ θα μπορούσε να αντιδραματίσει ένα ρόλο. Έχουμε επίση διαφορετικέ πρακτικέ στι διάφορε χώρε, οι οποίε συχνά παρεμποδίζουν τα διασυνοριακή εμπορία υπηρεσιών ακόμη και αν είναι κοινή η γλώσσα συνεννόησης. Και τι γίνεται με τις νέες υπηρεσίες που ακόμη δεν έχουν όνομα στι στις νέες τεχνολογίες, στην ε, ευημερία λόγου χάρη και την υγεία. Εδώ τι μπορεί να περιμένει κανείς εάν δεν έχουν συγκεκριμένο όνομα οι υπηρεσίες αυτές. Θα μπορούσε λοιπόν η τυποποίηση για να έχουμε μια κοινή συνεννόηση για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Θα πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη το πώς συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες στην Οδηγία 9834, μέρος του πακέτου τυποποίηση. Και θα πρέπει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ότι είναι τρέχουσα πρακτική των φορέων τυποποίηση και κατά πόσο θα κοινοποιούνται τα προγράμματά του. Ένα καθοριστικό σημείο είναι το να ευαισθητοποιήσουμε και να προωθήσουμε τα πλεονεκτήματα που μπορεί να ενέχουν τα πρότυπα για τι υπηρεσίε, αντιμετωπίζοντας και καλύπτοντα και κάποιε ανησυχίες που γίνονται καθημερινά. Ε, οι δημόσιε διαβουλεύσει για την τυποποίηση και το σχετικό πακέτο φαίνεται να στηρίζονται και δείχνουν στήριξη για την τυποποίηση στις υπηρεσίες. Όμως υπάρχουν και ενδιασμοί. Εδώ νομίζω υπάρχουν κυρίω τρει κατηγορίε ενδιασμών. Πρώτον, παρανόηση για τη διαδικασία, Κάποιοι νομίζουν δηλαδή ότι θα υπάρχει υπερβολική ενοποίηση και θα χαθεί η εξατομίκευση για τα τυποποιημένα παιχνίδια λόγου χάρη. Σαφώ και συνεχίζουν να υπάρχουν διαφορετικά αρκουδάκια όσο και αν είναι ίδια τα πρότυπα. Ε, έπειτα για την τυποποίηση, όταν αγοράζει κανεί ένα προϊόν, το κοιτάζει, το αγγίζει, μπορεί να το δοκιμάσει και μπορεί να το αφήσει πάλι στο ράφι, εάν δεν εκπληρώνει τι προσδοκίε του καταναλωτή. Αυτό πώ μπορεί να γίνει με μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται σε έναν πελάτη. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, όταν ε, κανεί οργανώνει μια έκθεση και πρέπει να πληρώσει του μεταφορεί, τι μεταφορικέ υπηρεσίε που θα φέρουν ε, λόγω χάρη εργατέχνη από όλο τον κόσμο. Εκεί θα θέλει κανεί να μπορεί να βεβαιωθεί ότι είναι μια η υπηρεσία που λαμβάνει λεγμένη, εξουσιοδοτημένη. Ότι η εταιρεία που προσλαμβάνει θα διαθέσει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τι ελεγμένε διαδικασίε. Μπορεί να μην είναι το μόνο σημαντικό κομμάτι, αλλά μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε επένδυση θα κάνουν εταιρείε. Και αυτό θα επηρεάσει και την αξία τους στην αγορά. Πρέπει εδώ επίσης να ενισχύσουμε την πολιτική και οικονομική στήριξη και να μην ξεχνάμε ότι τα ευρωπαϊκά υπηρεσιακά πρότυπα θα αναπτυχθούν και για εσωτερικούς σκοπούς, αλλά ενδεχομένως να αποτελέσουν και ένα μέτρο σύγκρισης για την διεθνή αγορά. Προχωρούμε όμως εδώ, έχουμε ήδη το σχετικό πρόγραμμα, έχουμε τη στρατηγική της ε, ευρωπαϊκής τυποποίησης για τις υπηρεσίες και επίσης για τις αεροπορικές και αεροπλοϊκές ε, υπηρεσίες που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σταθώ τώρα σε μια γενικότερη, στατικικότερη θεώρηση του θέματος και να αναφερθώ στη σημασία των διαπιστευμένων προτύπων υπηρεσιών για την τυποποίηση των υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προτύπων είναι αξιόπιστο διεθνώς και χρησιμοποιείται πολλές φορές για τα διεθνή πρότυπα είναι ένα ευρύτερο σύστημα του διεθνούς, του παγκόσμιου συστήματος. Στην Ευρώπη έχουμε ένα ενιαίο μοντέλο με πολύ συγκεκριμένε εμπειρογνωμοσύνε και πολύ καλή εναρμόνιση κανόνων. Πολλέ φορέ θεσπίζουμε ή συμπληρώνουμε ε, θεσμικούς ε, υποχρεωτικού κανόνες στα πλαίσια της καλύτερη νομοθεσίας. Αυτό γίνεται με τη χρήση τη ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και τη διάθεση ενίσχυση τη ευημερία στην Ευρώπη. Ευρώπη εννοούμε Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν, δηλαδή 31 χώρες συν 19 άλλες συνδεόμενες χώρες. Έτσι λοιπόν στην αναθεώρηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για αυτό το επιτυχημένο παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Συστήματο Τυποποίηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και του καθοριστικού παράγοντε επιτυχία του συστήματο, τι εθνικέ αντιπροσωπείε, την ουδετερότητα και ανεξαρτησία των παραγόντων που συμμετέχουν στο σύστημα, βεβαιωνόμενοι ότι κατά το σχεδιασμό των προτύπων δεν θα υπάρχει ένα ε, παράγοντα που θα υπερτερεί και θα υπερκεράσει του υπόλοιπου, και βεβαίω ότι όλα αυτά θα μπορούν να αξιοποιηθούν και στο διεθνέ ε, σύστημα τυποποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Να προσθέσω όσον αφορά το έργο της Επιτροπής πως ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τις διατάξεις της οδηγίας υπηρεσιών που ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να στηρίξουν προδιαγραφές για διασυνεργειακές υπηρεσίες και η κυρία Εύλιν Γκέπχαρτ αυτή τη στιγμή συντασμία έκθεση για την εφαρμογή αυτής της και νομίζω θα εξετάσουμε και αυτή τη πτυχή ταυτόχρονα οπότε νομίζω πως υπάρχει μια ευκαιρία εδώ πέρα να εξετάσουμε κάποιου από του παράγοντε που πολύ σωστά απεικονίσατε στην, έκθεση, στην παρουσίασή σα και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Περνάμε τώρα στι δημόσιε προμήθειε που είναι ένα εξίσου σημαντικό θέμα για αυτή την επιτροπή και ο κύριο Μάρκο Ράγκλ θα μα μιλήσει γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, όταν μου ζητήθηκε να συνεισφέρω για την χρήση προμηθειών, προμήθειες αναρωτήθηκα ποια είναι η διαφορά μεταξύ δημοσίων προμηθειών και μιας ιδιωτικής αγοράς, π.χ. μεταξύ δύο επιχειρήσεων. Και δεν υπάρχει καμία, μπορώ να σας πω. Και οι δημόσιες προμήθειες και οι ιδιωτικές στοχεύουν σε μια σύμβαση, τελικά σε μια συναλλαγή μέσω μιας σύμβαση και οι οικονομολόγοι, αν του ρωτήσετε, θα σπούν πούν πως ε, οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή αφορά τη μείωση της ε, συμμέτριας πληροφοριών, να μειωθεί το κόστος και ο ηθικός και τυχόν αποτυχία της λειτουργίας της αγοράς. Και για να διευκολυνθούν λοιπόν αυτές οι συναλλαγές μπορούμε να ρωτήσουμε γιατί μπορούν να βοηθήσουν οι προδιαγραφές. Πρώτα απ' όλα το να αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές ε, που αναφέρονται σε κάποιες οδηγίες σημαίνει πως υποθέτουμε πως υπάρχει συμμόρφωση στις ε, σχετικές νομικές απαιτήσεις. Οπότε υπάρχει ασφάλεια το ένα όφελος είναι αυτό. Δεύτερον, το αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές σημαίνει πως χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και πάντα έχουμε λύσεις σύγχρονες. Και βεβαίω βασιζόμαστε με το να αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε μια συνένεση μεταξύ όλων των ενδιαφέρον μερών που σημαίνει πως έχουμε συμπερίληψη όλων όσων έχουν συνεισφέρει μέσω των εθνικών αντιπροσωπείων. τρίτων το να χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές εξοικονομεί χρήματα και στην προκειμένη περίπτωση χρήματα των φορολογουμένων για το χαμηλότερο κόστος παραγωγής σημαίνει χαμηλότερη τιμή μέσω της εναρμονισμένης τεχνολογίας. Περισσότεροι πολιτές επίσης θα προσελκυστούν στον διαγωνισμό αυτό, θα ενταθεί ο ανταγωνισμός και άρα πάλι θα πέσει η τιμή. Και τέλος, θα έχουμε ευκολότερο τρόπο εξυπηρέτησης των προϊόντων και λύσεων που θα αγοράσει κανεί. οπότε μειώνεται εδώ πέρα το κόστος επισκευή και συντήρησης και άρα κύκλου ζωή. Οπότε, τέταρτον, το να χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ σημαίνει πω οι επενδύσει είναι πιο αηφόρες γιατί διασφαλίζεται διαλειτουργικότητα με την υπάρχουσα υποδομή, οπότε υπάρχει και μικρότερο κίνδυνο του να μην συμπληρωθεί, να μην ολοκληρωθεί ένα τυχόν έργο και οθεί τον ανταγωνισμό προς την καινοτομία και προς πιο καινοτόμα προϊόντα, άρα αυξάνεται η αποδοτικότητα των λύσεων που θα κανείς. Τούτων λεχθέντων τώρα θα ήθελα να καταλήξουμε το ερώτημα ποιο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης θα δώσει αυτά τα ωφέλη που θέλουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε, εάν θέλουμε, να έχουμε ασφάλεια μέσω της υπόθεσης συμμόρφωσης πρέπει να διατηρηθεί αυτό το μοντέλο το οποίο λέμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με εθελοντικές προδιαγραφές και εθελοντική συμμετοχή για να γίνει πιο συγκεκριμένος ε, η νομοθεσία η οποία αναφέρεται στις οδηγίες. Δεύτερον, εάν θέλουμε επίκαιρες και σύγχρονες λύσεις πρέπει να διατηρήσουμε την εθελοντική συμμετοχή στην διαδικασία τυποποίησης που βεβαίως ως κίνητρο θα έχει το συμφέρον και την σημασία μιας εταιρείας στην αγορά. Τέλος, εάν, τρίτον, εάν θέλουμε μια συνένεση και συμμετοχή όλων, πρέπει να ενισχύσουμε την αρχή των εθνικών αντιπροσωπιών και να ενισχύσουμε τους εθνικούς φορείς με τη δυνατότητα που έχουν να χαμηλώσουν τα εμπόδια συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων ε, χρηστών, καταναλωτών, ΜΚΟ, δημοσίων αρχών, βιομηχανίας και πολυεθνικών εκπροσώπων των εργαζομένων ε, της υγιεινής και ασφάλειας και των αναπήρων βεβαίως ως χρηστών των προϊόντων. Τέταρτον, εάν θέλουμε να εξοικονομήσουμε τα χρήματα των φορολογημένων μέσω του ανταγωνισμού πρέπει να ενισχύσουμε την χρήση προδιαγραφών στις δημόσιες προμήθειες μέσω της αύξησης ενημέρωσης των σχετικών φορέων που προκυρήσουν τις προμήθειες. Πέμπτον, εάν θέλουμε αηφόρες λύσεις στις δημόσιες προμήθειες μέσω της διαλειτουργικότητας πρέπει να διαφυλάξουμε την ακαιρεότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης και την συνοχή των παραδοτέων, δηλαδή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτό μπορεί να γίνει με το να επαναληφθεί η γνωστή αυτή ομάδα Sensenelec και έτσι, σύμφωνα με την οδηγια 9834, ενώ μπορούμε μέσω της ε, μεθοδολογίας να οδηγηθούμε σε παραδοτέα για την λεγόμενη μη πλήρη συνένεση, όπως παραδείγματο χάρη οι φόροι και γινοπραξίες εντός του υπάρχοντος συστήματος. Τώρα να σας πω κάποια καλά νέα από τη γερμανική βιομηχανία, την οποία εκπροσωπώ εδώ πέρα τα βιβλία παραγγελιών μας πάλι γεμίζουν για μεγάλο κομμάτι της γερμανικής βιομηχανίας, ειδικά όσον αφορά το βιομηχανικό τομέα και το κατασκευαστικό τομέα. Η οικονομική κρίση τελείωσε, η ατμομηχανή ξαναπαίρνει προς και στη σωστή, βρίσκεται στη σωστή πορεία και όλοι ξέρουμε βεβαίως πως πρέπει να σύρει πολλά βαγόνια. Αλλά θα πρέπει να θυμάστε πως η γερμανική βιομηχανία δεν είναι μόνο η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης είναι και η ατμομηχανή τυποποίησης και ε, όταν μιλάω για τη γερμανική βιομηχανία ε, εννοώ και τις μεγάλες βιομηχανίες και τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις βεβαίως και ένα από τα μέσα για να συνεχίσει να λειτουργεί η ατμομηχανή ένα αρκετά σημαντικό θα έλεγα είναι να λειτουργεί σωστά το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης. Νομίζω πως όλοι ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κοινό. Thank you. Uh, thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ράιγκλ. Ελπίζουμε η αισιοδοξία σας για τις μελλοντικέ εξελίξεις στην παραγωγή σε όλη την Ευρώπη να γίνουν πραγματικότητα. Και τώρα θα, ρωτήσω, θα ζητήσω τον κύριο Φρίντριχ να μας πει κάποια λόγια για κάποια τεχνικά ζητήματα, γιατί είναι μέρος ε, του πάνελ των εμπειρογνωμόνων και ασχολείται με την τυποποίηση των ε, τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση να με σας μιλήσω σήμερα. Όπως ταξίδευα χθε από τη Χαϊδελβέργη, την πόλη μου, Πήρα το τρένο ως συνήθω και προσπάθησα με αυτή την ωραία εικόνα να σας δείξω πώς είχαν τα πράγματα. Πολύ άνετα ήταν στο τρένο, είχα το λάπτοπ μου, Εκεί λειτουργούσε σύστημα, λειτουργούσαν όλα τα και το σύστημα Wi-Fi ασύρματη σύνδεση. Και έπειτα μπορούσα να παρακολουθήσω τις πρόσφατες ειδήσει, να δω την σελίδα της εταιρεία μου μέσω του ιδιωτικού μα κλειστού δικτύου, μπορούσα να δω και το email μου. Είχα πολλά μηνύματα χθε. Ευτυχώ γιατί έλαβα πολλά και πρόσω... κατάφερα πολλά να κάνω στο ταξίδι για Βρυξέλλες. Και μετά έκανα και κάποια δουλειά, δηλαδή αντάλλαξα κάποια έγγραφα με του συναδέλφου, έγγραφα που είχαμε να ετοιμάσουμε και που δεν είχα προλάβει να κάνω νωρίτερα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη χρήση προτύπων Αυτές ε, οι τεχνολογίες χρησιμοποιούν τα πρότυπα ICT, διεθνή πρότυπα ICT. Νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην αίθουσα αυτή χρησιμοποιούν το ίδιο είδος τεχνολογιών και το ίδιο, το ίδιο είδος προτύπων. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε μια πολύ μικρή συνοπτική εικόνα της τυπικής εικόνας των ποιο είναι τα διεθνή πρότυπα Αν δούμε την δεξιά κολόνα του οργανισμού θα δείτε από πού προέρχονται. Από την ITF, από την W3C, από την ISO, το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που ετοιμάζουν πρότυπα. Αυτό όμως που είναι σαφές είναι ότι καινοτόμες τεχνολογίες ICT συνδυάζουν διαφορετικά πρότυπα από διαφορετικά είδη οργανισμών. Εδώ βλέπετε επίσης μια συνοπτική εικόνα του διεθνούς οικοσυστήματος τυποποίησης ICT. Στην πρώτη γραμμή, την κόκκινη γραμμή με τις τελείες, βλέπετε τους πυλώνες των φορέων που είναι αναγνωρισμένοι για την τυποποίηση διεθνώς. Το W3C, την OASIS και ούτω καθεξής. Όλα αυτά καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης σήμερα. Από την Οδηγία 9834. Στο επόμενο σημείο της διαφάνειας, μεταξύ των δύο διακεκομένων κόκκινων γραμμών, βλέπετε τους οργανισμούς κοινοπραξίες και φορά που αναφέρονται, που είναι ανεπίσημοι φορείς τυποποίησης. Είναι προμηθευτές προτύπων ICT, δεν είναι επισήμως αναγνωρισμένοι και βρίσκονται εκτός του πεδίου της ευρωπαϊκής τυποποίησης του σχετικού πλαισίου σήμερα. Άρα τα πρότυπα από τους οργανισμούς αυτούς δεν διατίθενται ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στους δημόσιες προμήθειες. Όπως είπα όμως νωρίτερα όλοι τα χρησιμοποιούμε και οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν με τρόπο ανοιχτό και διαφανή χρησιμοποιούν μια σειρά από κριτήρια, έχουν υλοποιήσει τις ε, διαδικασίες ICT, μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν σε αυτά από όλο τον κόσμο. Γενικώ έχουν διεθνή εμβέλεια λόγω της διεθνούς διάστασης των ε, τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Και βλέπετε και την επόμενη διακεκομένη κόκκινη γραμμή. Εκεί έχετε τα κλειστά φόρα και κοινοπραξίες Ιδιωτικού φορείς, ας πούμε. Εμείς μιλάμε όμως κυρίως για τη μεσαία ζώνη, του οργανισμού που βρίσκονται στη μέση. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα. Ένα μεγάλο μέρος της τυποποίηση ICT γίνεται από οργανισμούς διεθνεί, ανοιχτού, εκτός όμως του σημερινού πλαισίου της ευρωπαϊκής τυποποίηση. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη μεταρρύθμισης εδώ. Οι τεχνολογίε επικοινωνία και πληροφορίας σε πολλές μελέτε έχουν εντοπιστεί, αλλά και σε διαβουλεύσεις και σε επιτροπέ εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εντοπιστεί ω ο τομέα, όπου η μεταρρύθμιση απαιτείται κατεπηγόντω. Τα διεθνή πρότυπα ICT από διάφορα φόρα και κοινοπραξίε είναι απαραίτητα για την κοινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Δείτε για παράδειγμα το διαδίκτυο, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως για την ιστορία μου με το τρένο, ή ε, και την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική ενέργεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το έξυπνο δίκτυο, ε, το cloud computing, πολλοί από αυτού του τομεί αναφέρονται ω ιδιαίτερα καινοτόμοι, προοδευτικοί τομεί σήμερα. Μπορεί να αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο η Ευρώπη, αλλά κανένα δεν θα φέρει τα απαιτούμενα αποτελέσματα χωρί να συμπεριλάβουμε τα διεθνή πρότυπα ICT των ε, ανοιχτών αυτών κοινοπραξιών και φόρων που σα ανέφερα. Η ψηφιακή ατζέντα που πρόσφατα δημοσίευσε η Επίτροπο Κρού είναι αναπόσπαστο μέρο τη στρατηγική Ευρώπη για το 2020. Έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο διεθνώ στι τεχνολογίε ICT και στο πόσο ανοιχτέ θα είναι αυτέ οι τεχνολογίε. Όμω όλα αυτά εξαρτώνται κατά πολύ από τα συγκεκριμένα πρότυπα, από τα διάφορα φόρα και κοινοπραξίε των τομέα των τεχνολογιών επικοινωνία και πληροφορία. Εδώ προτείνεται Υπάρχει μια λύση που προτείνεται από καιρό, εξετάζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανέφερε, την ανέφερε στην ομιλία της το πρωί. Το 2006 η Επιτροπή ξεκίνησε με μια μελέτη ICT και τα αποτελέσματα συνοψίστηκαν σε μια διάσκεψη πάλι με ένα έγγραφο που συνόψιζε τα πορίσματα της Επιτροπής και τελικά με συγκεκριμένες προτάσεις στη Λευκή βίβλο τη Επιτροπής για τον εξυγχρονισμό των προτύπων ICT για την Ευρώπη. Οι δημόσιε διαβουλεύσει έχουν ολοκληρωθεί, είχαν τεράστια στήριξη και επίση από ολόκληρο τον κλάδο των ICT στην Ευρώπη. Η μελέτη αντικτύπου έχει ολοκληρωθεί και τα πάντα είναι έτοιμα. Η πρόταση είναι να αναθεωρηθεί η απόφαση του Συμβουλίου 8795 η απόφαση αυτή του Συμβουλίου επικεντρώνεται στη χρήση και την εφαρμογή των προτύπων στον τομέα ICT για να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα. Προτείνει επίση να υλοποιηθούν διαδικασίε για να χρησιμοποιηθούν διεθνή πρότυπα ICT στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και τι δημόσιε προμήθειε, λαμβάνοντα υπόψη τα κριτήρια του κατά πόσο πρέπει να είναι ε, δυνατή η πρόσβαση, των απαιτήσεων επίση ε, συμμόρφωση των ευρωπαϊκών προτύπων. Η προτινόμενη λύση που και ο βιομηχανικό κλάδο ε, προάγει είναι η αποσύζευξη των προτύπων αυτού, αυτών από το πεδίο της οδηγίας. Ας δούμε και την επόμενη διαφάνεια, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση ICT. Τα διεθνή πρότυπα λοιπόν ICT είναι κρίσιμη σημασία για την Ευρώπη, ώστε να αναλάβουμε εδώ για την ρόλο στην κοινοτομία. Μία πλήρης ε, αντισύλληψη του θέματος για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ICT και της πολιτικής τυποποίησης έχει αναπτυχθεί με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Και θα πρέπει να έχουμε το απαραίτητο πλαίσιο για τη χρήση των διεθνών ε, προτύπων ICT που να είναι, ε, να είναι διεθνής, διεθνούς εμβέλειας και να υπάρξει και αποσύζευξη από το πεδίο της οδηγίας 8934 κατά τη μεταρρύθμισή της. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πολύ σαφή παρουσίαση. Να περάσουμε τώρα στο τελικό μέρος των ερωτήσεων. Έχω εννέα συναδελφούς που έχουν ζητήσει το λόγο και μετά θέλω να δώσω και το λόγο στους ομιλητές μας. Θα σας δώσω λοιπόν από ένα λεπτό και ας προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Πέντε οι ομιλητές, ας ακούσουμε λοιπόν τους πέντε ομιλητές και θα δούμε πώς χρειαστούν και οι ομιλητές από τα προηγούμενα πάνε λίγο χρόνο για να απαντήσουν. Μπορεί να θέλετε να πείτε κάτι που ξεχάσατε σαν έναν από τους πρώτους παρεμβαίνοντες. Εάν έχετε λοιπόν κάποιο σχόλιο να κάνετε, παρακαλώ να μου το επισημάνετε. Επίσης ακούσαμε από την Κομισιόν, δεν ξέρω αν η κυρία Βάισμαν παρούσα και αν θέλει να λάβει το λόγο σήμερα, αλλά σίγουρα θα έχει την ευκαιρία να παρέμβει εφόσον το επιθυμεί. Θα σας δωσω δυο δύο-τρία λεπτά. Φυσικά πάντα θα συμβάλλετε και στην εκπόνηση της εκθεσή μας. Λοιπόν, να σας πω ποιοι είναι οι ομιλητές, οι ισχυώδεις εισηγητές και οι συντάκτες νομοδότησης, ο κύριος ε, Κόζισνικ, Μπουτικόφερ Κόνι, Ρέφερ, Ρούλα, Βάιλερ και Κορία. Ένα λεπτό, ο καθένας σας, ο κύριος εισηγητής, κύριο Κούζεσνικ. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Την προηγούμενη εβδομάδα συνάντησα τον κύριο Γιάννη από την ΟΡΠΑΠΜΕ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή του για την έκπτωση που θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις συστάσεις του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό ποιος θα καταβάλει το κόστος αυτό που θα προκύψει από την έκπτωση, αυτό το πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, ίσως, για το δεύτερο μπορώ να επανέλθω αργότερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ κύριε Μπίτι Κόφερ. Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα. Ένα για τον κύριο Κουτσογιάννη. Μάλλον συνδέεται με τον κύριο Κουτσογιάννη, αλλά έχει να κάνει και με άλλους ομιλητές. Κύριε Κουτσογιάννη, μιλήσατε για την ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την θεσμική τους αναγνώριση, institutional recognition. Θα ήθελα να ρωτήσω τα άλλα μέλη των πάνελ που έχουν ε, αναφερθεί υπέρ της ανάγκης εθνικής εκπροσώπησης, αν συμφωνούν για αυτή την πρόταση ή που πρέπει να την περιορίσουν, εάν όχι απόλυτα. Για τον κύριο Χάρης επίσης, αν σας κατάλαβα καλά, είπατε ότι οι διαδικασίες τυποποίησης και στο μέλλον θα πρέπει να εστιάσουν στα προϊόντα και οι προκλήσεις της κοινωνίας δεν μπορούν να καλυφθούν με τη μέθοδο της τυποποίησης, αλλά θα πρέπει να, κατα... να καλυφθούν από μια νομοθετική διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια επιχειρηματική κοινότητα να μιλάει για περισσότερη νομοθεσία. Θα ήθελα να ξέρω κύριε Χάρης αν μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα για κάποιες προκλήσεις κοινωνικές που κατά την άποψή σας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ή δεν έχουν αντιμετωπιστεί με την τυποποίηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε τι γίνεται με τι 58 συστάσεις τη Σανελέ και της για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχουν και διεθνεί μελέτε που δείχνουν ότι παρέχει πολλέ δυνατότητε η δική του συμμετοχή στην όλη διαδικασία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώ και οι ίδιε οι συστάσει. Όμω ακόμη δεν είμαστε σε θέση να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη εδώ. Η έκθεση Μόντι έδειχνε την ανάγκη να δημιουργηθεί επιχειρηματική, επιχειρηματικό περιβάλλον πιο αρμονικό και ευνοϊκό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να μπορέσουν να υποφεληθούν από τα πλεονεκτήματα όλου αυτού του συστήματο. Ο στόχο εδώ προφανώ είναι να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και την εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οπότε, εδώ έρχεται και το έτοιμά μου. Κάποιοι από εσά σε διάφορε συναντήσει είπαν ότι τα πρότυπα μπορούν να διαφέρουν στου διάφορου τομεί και είσαστε κατά τη ε, ρύθμιση που μπορεί να είναι κατακαιρματισμένη ή θέλετε μια τυποποίηση ενοποιημένη και να εκπροσωπεί όλε τι διαφορετικέ περιπτώσει μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο κύριος Μπράντεν και άλλοι αναφερθήκαν ήδη στο θέμα αυτό ότι θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια να προωθηθούν τα πρότυπα διότι τα πρότυπα και να γίνουν πιο κατανοητά. Δεν ξέρω μας αν ζούμε στον ίδιο κόσμο. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα πρότυπα είναι ένα πρότυπο ακόμα και εάν οδηγούν και σε κάποιες προκλήσεις. Το ερώτημά μου λοιπόν θα ήταν το εξής. Κατά πόσο έχει μελετηθεί σε βάθος η βασική φιλοσοφία του συστήματος τυποποίησης. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει εξ αρχής, θα πρέπει να προβλέψουμε μια οδηγούσα φιλοσοφία τυποποίησης, παραδείγματος χάρη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των τεχνικών και των μηχανολόγων. Γιατί θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να υπάρχουν κάποιε βασικέ προδιαγραφέ οι οποίε θα είναι χρήσιμε και για αυτού και χρήσιμε και για του καταναλωτέ. Υπάρχει επίση και η ανάγκη να έχουμε κανόνε για την ανθρώπινη ευμάρεια. Και έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημά μου. Τι προβλέπετε για την τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών, για ποιε τυποποίησει μιλάτε, για ποια πρότυπα και σε ποιο βαθμό. Η κυρία Ρούλα. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις έχω προς την κυρία Μπλάχα. Είπατε πως οι εθνικές αντιπροσωπείες πρέπει να διασφαλίσουν πως υπάρχει δημοκρατική νομοποίηση, αλλά ακούσαμε τώρα πως οι ενδιαφερόμενοι είναι διαφορετικοί στα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη δεν ε, έχουν αρκετή εκπροσώπηση των επιχειρήσεων. Τι θα κάνατε εσείς και κατόπιν μιλήσατε για τον τρομέα των υπηρεσιών, αλλά ακούσαμε από τον τομέα επικοινωνίας και προφορικής πως θέλουν μια διαφορετική βάση. Θεωρείτε πως είναι η ίδια η νομική βάση για αγαθά και υπηρεσίες και τέλος ε, για τις δημόσιες προμήθειες. Εντάξει, ωραία τα πράγματα με τις προδιαγραφές, αλλά εγώ έχω την εμπειρία ε, όπου στο Fair Trade που είναι εθελοντικές προδιαγραφές δεν τις αναγνωρίζει αυτές η Κομισιόν ή αν θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια συμπεφωνημένα πρότυπα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει αντιμετωπιστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξάλλου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βάιλα. Και εγώ αναρωτήθηκα για αυτό που είπε ο εκπρόσωπος των γερμανικών ενώσεων δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά Είπατε ότι όλα πάνε πολύ καλά, ότι λειτουργεί πολύ καλά και ανθεί το επιχειρηματικό κλίμα, ενώ από την άλλη πλευρά ελέγχθη από τους άλλους ομιλητές ότι υπάρχει μια ανάγκη μεταρρύθμισης, ιδίως στον τομέα των ε, νέων τεχνολογιών. Και έρχομαι και σε αυτά που είπε ο κύριος Κουτσογιάννης, ότι πολλές φορές τα πράγματα γίνονται σε ένα κλειστό κύκλωμα και είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει μια συμμετοχή σε επίπεδο εμπειρογνωμών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα πιστεύω ότι αυτή η ακρόαση θα πρέπει να βοηθήσει ώστε ο εισηγητής μας να μπορέσει να καταλήξει και σε κάποια σύνοψη προτάσεων προς την Κομισιόν, γενικά προς τους νομοθέτες εμείς λοιπόν μας ενδιαφέρει να ξέρουμε για το αν πηγαίνουν τα πράγματα όλα θαυμάσια στον αγγελικό αυτό κόσμο ή αν υπάρχουν οι δυσκολίες αυτές για πρόσβαση στις πληροφορίες. Για τις υπηρεσίες τέλος πιστεύω ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Γερμανίας υπάρχουν ορισμένες ε, υπηρεσίες οι οποίες την χάνουν μιας προτυποποίησης, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν και επομένως, παραδείγματος για ορισμένα είδη περίθαλψης και φροντίδας, χρειάζεται να υπάρχει αυτή η τυποποίηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια αντίστοιχη ε, πρόβλεψη για άλλους, ε, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ίσως θα μπορούσε να μας το πει αυτό ο εκπρόσωπος των γερμανικών φορέων, Μήπως αυτό θα μπορούσε να δώσει μια δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν τις υπηρεσίες φροντίδας και περίθαλψης τις οποίες μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν και ποιες όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουρία Ντικάμψου. Η ερώτησή μου αφορά τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες ή procurement. Άκουσα την παρέμβαση του κ. Ράγκλ για τις δημόσιες προμήθειες με προσοχή και τα πρότυπά του και παραξενεύτηκα που δεν έγινε μια ιδιαίτερη μνήμα για τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. Εδώ σημαίνει ότι θα υπάρχουν πλατφόρμε μεταξύ του αυτού που έχει προκηρύξει το διαγωνισμό και του υποψηφίου αλλά αυτές οι πλατφόρμες δεν διατίθενται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό αυτό στα πλαίσια του e-procurement. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί ευκαιρία αυτές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και να ωφελήσει για την εισαγωγή των προτύπων και των προδιαγραφών. Υπάρχει σίγουρα μέρημνα για τις μεγάλες εταιρείες, αλλά το e-procurement και σχετικέ πλατφόρμες θα πρέπει να είναι μια αξία που όλοι θα μπορούν να εκμεταλλευτούν. Um, Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε πάλι να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Φρίντριχ ως πρόεδρος για την πρότασή του την οποία θα ήθελα να διευκρινίσει. Από ό,τι κατάλαβα από τις συζητήσεις μας σήμερα το θέμα της συμπερίληψης αυτών των ειδικών ομάδων πληροφορικής στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης νομίζω πράγματι το στηρίζουν όλοι για την επίτευξη των στόχων. Οπότε δεν ξέρω γιατί πρέπει να αποσυνδεθεί εφόσον προς αυτή την κατεύθυνση πάμε. Εάν ζήτω για κάποια συγκεκριμένη στήριξη για την υιοθέτηση αυτών των προδιαγραφών θα ήταν εκτός του θέμα της σημερινής συζήτησης, αλλά δεν νομίζω ότι τα δύο ε, είναι ασύμβατα υπ' αυτή την έννοια. Οπότε νομίζω πως σήμερα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι θέλει, εάν θέλετε, η ε, κοινότητα πληροφορικής και επικοινωνιών από το ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, εντάξει, μπορεί να θέλει διαφορετικά πράγματα από τη χρήση, αλλά εδώ πρέπει να λέμε για την ανάπτυξη των προδιαγραφών. Οπότε θα ήθελα να τώρα να ζητήσω από τους πέντε ομιλητές μας να απαντήσουν. Θα σας δώσουμε από ένα λεπτάκι γιατί πρέπει να τελειώσουμε όλα. Έντριαν Χάρης λοιπόν πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω πρώτα απ' όλα την ερώτηση του κύριου Μπιτικόφερ. Για μας είναι σαφές πως οι ρυθμιστικές αρχές θα ορίσουν ποιο είναι το βασικό νομικό πλαίσιο στην, είτε στην υγιεινή και ασφάλεια περιβάλλον, είτε στο πώς συμπεριφέρονται οι εταιρείε. Αυτό το ορίζει η ρυθμιστική αρχή. Και μετά η τυποποίηση είναι ένα εργαλείο για να μεταφραστεί σε προϊόν η υπηρεσία. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι μια τάση έτσι, φέρπουσα να πηγαίνουν οι εντολές τυποποίησης πέρα από τις απαιτήσει του νόμου και να συμπεριλαμβάνουν κάποιες άλλες πολιτικές επιλογές που παρακάμπτουν την κανονική νομοθετική διαδικασία. Για να επανέλθω όλο το ερώτημα που έγινε για την αρχή των εθνικών αντιπροσωπείων. Είναι σαφές πως η τυποποίηση είναι δημοκρατική διαδικασία. Λειτουργεί καλύτερα όσο πιο κοντά είναι στους ενδιαφερόμενους. Γι' αυτό λέμε πως είναι σημαντική η αρχή των εθνικών αντιπροσωπείων γιατί εκεί μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι Βρυξέλλες είναι πολύ μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να το θυμάστε αυτό. Ευχαριστώ ο κύριος Γκουτσογιάννης για το θέμα τώρα του ποιος πληρώνει για την έκπτωση στις προδιαγραφές για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις σε περίπτωση που μια εθνική κυβέρνηση αποφασίσει πως θέλει κάποιες προδιαγραφές να είναι δωρεάν πρέπει βεβαίως να αποζημιώσουν τους οργανισμούς που χάνουν αλλά η πρόταση που κάνουμε για ειδικέ εκπτώσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει άλλο νόημα. Σήμερα με τους υπολογισμούς μας μία στι πέντε εταιρείε αγοράζει ένα πρότυπο το έτος. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρεών δεν αγοράζουν ποτέ προδιαγραφές. Εδώ πέρα λοιπόν δεν έχουμε στόχο να μειώσουμε τα έσοδα των ε, οργανισμών προδιαγραφών, αλλά να τα αυξήσουν με το να αποκτήσουν νέου πελάτε στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Οπότε δεν χρειάζεται αποσμίωση. Για το εάν τώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν η τυποποίησή τους πρέπει να γίνει γενική, όχι, πρέπει να γίνει ανατομής, αλλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι γενική ενθάρρυνση και στήριξη ίσως τεχνική και οικονομική για να συμμετάσχουν και αυτές οι εταιρείες στην σύνταξη π.χ. τομεακών προδιαγραφών και έγινε μια ερώτηση για το αν είναι εύκολη διαθέσιμη πληροφόρηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει καταγραφεί ότι δεν το θεωρούν αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εμείς έχουμε την εντύπωση πως είναι υπόθεση ε, εμπειρογνωμόνων να προσπαθήσουν να βρουν τη σωστή προδιαγραφή έτσι όπως γίνουν τα πράγματα σήμερα. Αυτό πρέπει να αλλάξει και ευτυχώς υπάρχει ένα καλό σχέδιο για να γίνει αυτό. Κύριε Μπλάουγκα, εγώ είδα έξι ερωτήματα που αναφέρονται σε μένα. Θα είμαι να τον πιο σύντομη. Καταρχήν αυτά που είπε ο κ. Κουσούσνικ. Ζητάτε να υπάρξει υποστήριξη για την ευρύτερη ε, διάδοση των standards και στη δική μας χώρα έχουμε συμφωνίες με τις ενώσεις αυτές για μια μεγαλύτερη ε, διάδοση και μας ενδιαφέρει λοιπόν να υπάρχει μια ευρύτερη διάδοση, αλλά μπορεί να γίνει αυτό με ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για αυτά που είπε ο κ. Μπιτικόφερ, για την θεσμική αναγνώριση. Έχουμε θεσμική αναγνώριση, όπως συνορπάπουμε και άλλοι φορείς που αναγνωρίζονται. Και έχουμε πολλούς εταίρους στο σύστημά μας, αλλά αυτό δεν επιλύει το θέμα της εμπειρογνωσύνης που πρέπει να υπάρχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκεί χρειάζεται υποστήριξη. Τρίτο σημείο, η τυποποίηση των υπηρεσιών σας. Παραπέμπω στο λεγόμενο πρόγραμμα CHESS, το οποίο ανέπτυξε η ΣΕΝ. Θα χρειαζόταν πολλοί χρόνο για να σα δώσω όλε τι λεπτομέρειε, αλλά μπορούμε στη συνέχεια να σα δώσουμε περισσότερη πληροφορία για το θέμα αυτό. Τέταρτο ερώτημα. Διαφορές στις πραγματικότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εθνικές αντιπροσωπείες. Εμείς πάντα Έχουμε φυσικά διαφορετικές καταστάσεις που ισχύουν στις χώρες μας και εδώ το πρόγραμμα της ε, μεταλαμβάνευσης βελτιστής των πρακτικών και ε, αξιολόγησης από μοτίμους της ΕΝΕΛΕΚ μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να ενισχυθούμε από τις επιτυχίες και να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις επιτυχίες που έχουν κτηθεί και όχι στα προβλήματα μονάχα. Πέμπτο ερώτημα αν πρέπει να υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις χωριστές για τα προϊόντα, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τεχνολογιών, ICT παραδείγματος χάρη, δεν μπορείτε να υπάρξει απόλυτος διαχωρισμός για θέματα συντήρησης. Επίσης, με την τεχνολογική σύγκληση, εγώ δεν βλέπω γιατί αυτοί οι τρεις τομείς θα πρέπει να είναι και χωρισμένοι. Τελευταίο σημείο, η σημασία της πιστοποίησης για την προώθηση των προτύπων. Ναι, όταν κανείς είναι υπεύθυνο για την αγορά υπηρεσιών για μια εταιρεία ή για τον εαυτό του. Είναι πολύ καλή η πιστοποίηση αυτή, δίνει όλο και περισσότερε κατευθύνσει. Όλο και περισσότερε εταιρείε χρησιμοποιούν την πιστοποίηση σαν ένα φίλτρο για να δείξουν ότι μπορούν πράγματι να είναι αξιόπιστοι στι υπηρεσίε και τα προϊόντα. Κύριο Ράγκελ. Και εγώ θα ήθελα να έρθω στο ερώτημα το οποίο συζητήθηκε ήδη για την εθνική εκπροσώπηση των πιο ασθενών ομάδων συμφερόντων τους έναντι υπερεθνικών δομών που θα πρέπει να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Πιστεύουμε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη Γερμανία, ότι η συμπερίληψη των συμφερόντων των πιο ασθενών ομάδων εμπλεκομένων μπορεί να γίνει με τον καλύτερο τρόπο σε τοπικό επίπεδο. Εκεί που είναι οι επιχειρήσεις, εκεί που ζουν τα άτομα αυτά, εκεί που βρίσκεται η, ο φυσιολογικός χώρος εγκατάστασης αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να έχουν από γεωγραφική αλλά και πολιτιστική έποψη μια πολύ μικρή απόσταση να διατρέξουν για να φτάσουν στον εθνικό φορέα προτύπων, ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να συμβάλλουν στη διαδικασία τυποποίησης. Αλλά δεν θα ήταν κακό να υπάρξει αυτή η εκπροσώπηση και σε υπερεθνικό επίπεδο, όπως παραγωγής χάρη όπως είπε ο κύριος Ράσελ, για τους καταναλωτές, για το περιβάλλον, όπως είπε ο η άποψή μας παραμένει ότι μια τέτοια υπερεθνική εκπροσώπηση, η οποία θα είναι θεσμοποιημένη σε φορείς όπως αυτούς που ανέφερα προηγουμένως, πιστεύουμε ότι αντί να διεκδικηθεί απλώς η εκπροσώπηση αυτών των ομάδων, θα πρέπει να δοθεί συγχρόνως και μια υποστήριξη προς τι εθνικές αντιπροσωπείες στις μικρότερες χώρες για να μειώσουν το, το άχθος της συμμετοχής των μικρότερων εμπλεκομένων. Και δεν υπάρχει έλλειψη υποδειγμάτων για να τα πετύχουμε αυτά, να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των μικρομεσαίων ε, εμπλεκομένων. Αυτά τα μοντέλα λοιπόν μπορούν να περάσουν από τη μία χώρα στην άλλη, να θεωρηθούν ότι είναι μια βέλτιστη πρακτική και να χρησιμοποιηθούν και στα νέα κρατημέλη. Ώστε να μπορέσουν οι χώρες αυτές να έχουν και κάποια μεγαλύτερη βοήθεια για να βελτιώσουν την διαχείρισή τους για πιο περιεκτικές διαδικασίες. Για την ηλεκτρονική προμήθεια, όπως ε, ζητήθηκε από τον κύριο Κορέα Ντεκάμπους. Δεν ξέρω ποιε είναι οι δυσκολίε που θα αντιμετωπίσουν οι μικρότερε επιχειρήσει οι οποίε συμμετέχουν στι ηλεκτρονικέ προμήθειε, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να υπάρχουν πραγματιστικέ λύσει χάρη στι διαδικτυακέ τεχνολογίε για να μειώσουμε και το φράγμα αυτό για τι μικρότερε εταιρείε. Ευχαριστώ. Και τέλο ο κύριο Φρίντριχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομα για το ζήτημα των ηλεκτρονικών προμηθειών αναφέρω το έργο Pebble, το οποίο μπορεί να το ξέρουν κάποιοι ε, πολλά μέλη αναπτύσσουν μια πλατφόρμα δημοσίων προμηθειών που βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα πληροφορικής και αν συμβεί κάτι τέτοιο τα εμπόδια για μικρομισές επιχειρήσεις ή οποιονδήποτε για να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες θα είναι πολύ χαμηλά. Και έρχομαι άρα εδώ πέρα στο δεύτερο σημείο, συμφωνώ με τον κύριο Ράγκελ πως είναι σημαντικές οι προδιαγραφές για τις δημόσιες προμήθειες και αν οι προδιαγραφές αυτές είναι ανοιχτές, αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα, γιατί έτσι μπορούν διάφοροι ανταγωνιστές να προσφέρουν τα προϊόντα τους όταν αναπτύσσουν ε, προδιαγραφές. Ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας τρίτων. Γιατί υπάρχει ανάγκη μεταρρύθμισης της τυποποίησης ε, των τεχνολογιών Ιστή. Αυτό χρειάζεται κυρίως στον τομέα της άσκησης πολιτικής. Αν θέλουμε να έχουμε πολιτική καινοτομία, θέλουμε να αναφέρουμε τις σημαντικές παγκόσμιες προτεγραφές, το wireless LAN που ανέφερα ή οτιδήποτε, τις προτεγραφές του διαδικτύου. Αν θέλουμε να προωθήσουμε τους έξυπνους μετρητές, ε, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάποιες αναφορές, κάποιες παραπομπές. Επίσης, ε, για να εφαρμόσουμε την πλατφόρμα αυτή προμηθειών που ανέφερα. Αυτή είναι η ανάγκη. Και η ανάγκη είναι η χρήση των προδιαγραφών για να επιτευχθεί και να προωθεί η διαλειτουργικότητα. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό από την Οδηγία 9834 που καλύπτει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών για μια εναρμονισμένη αγορά που στηρίζει την ρύθμιση. Γι' αυτό πιστεύουμε πως στον τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών το παρελθόν η οδηγία 87-95 λειτουργούσε μια χαρά και το να υπάρχει μια ειδική οδηγία για αυτόν τον τομέα χρειάζεται. Γι' αυτό θεωρούμε πως χρειάζεται μια αναθεώρηση αυτής της απόφασης ε, για να καλύψουν τομέα ICT και δεν χρειάζεται ξανά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ και θεωρώ πως πρέπει να συγκεκριτήσουμε και για αυτά τα οποία μας είπατε τώρα. Now Λοιπόν. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας σχεδόν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κουζουνιέκ για να μας πει τι θα κάνουμε στο μέλλον. Αλλά θα ήθελα να δώσω και στην κυρία Ρενάτε Βάισενχόρν, η οποία είναι η επικεφαλής αντίστοιχης μονάδος τυποποίησης στην Κομισιόν, να μας πει δύο λόγια. Θα έχουμε φυσικά την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε στα πλαίσια της εκθέσης του κ. Κουσουσνίκ, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε και τα λόγια σας. Στο λόγο στο Ματία Πελεγκρίνη, ο οποίος θα μιλήσει εξ ονοματός μου. Και εγώ θα επανέλθω βέβαια. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που είχαμε αυτή τη γενική συζήτηση, καθότι βρισκόμαστε πρώτων πυλών της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου δεν είναι καινούριο και φαίνεται γενικώ αποδεκτό ότι η τυποποίηση μπορεί να επηρεάζει και τη μεταφορά τεχνολογιών και θα πρέπει να ξαναδούμε την αλληλεξάρτηση τυποποίηση και έρευνα. Χαίρομαι που αυτό είναι ευρέω πλέον αναγνωριζόμενο, αλλά είναι και σημαντικό για το μέλλον τη τυποποίηση. Σα διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στην ε, τρέχουσα αναθεώρηση και το σύστημα αυτό ήδη λειτουργεί ομαλά, όμως οι σημερινές μας συζητήσεις έδειξαν ότι υπάρχουν ακόμη πολλές ανάγκες και κυρίως η ανάγκη να συζητήσουμε περαιτέρω, να υπάρξει διάλογος. Χρειάζεται λοιπόν και άλλος διάλογος και ίσως και τεχνικότερος μακροπρόθεσμα. Δεν μπορούμε να βρούμε μόνο έναν τρόπο για τις ε, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και τις νέες τεχνολογίες και να τα συνδυάσουμε με έναν μόνο τρόπο όμως πολύ ευπρόσδεκτες ήταν οι ιδέες όλων των ε, παρεμβενόντων και σίγουρα υπάρχει ένας νέος ε, δρόμος πάνω για την τυποποίηση, νέα παιδεία και αυτό θα μας ε, θα φανεί και μέσα από τις μελλοντικές συζητήσεις μας για το θέμα. Ε, ευχαριστώ. Είμαι και εγώ μέλος του επιτελείου του κυρίου Ταγιάννη για τα θέματα τυποποίησης. Ξέρετε ότι είναι στη Νέα Υόρκη, εκείνος, όμως εγώ η Σίλβια και άλλοι συνάδελφοι από το επιτελείο έχουμε παραμείνει στο τέλος της ακρόασης. Η αξία τη τυποποίηση μεταξύ τη χθεσινή ημέρα και σημερινή ε, επιβεβαιώθηκε νομίζω γιατί χθε είχαμε την συνεδρίαση τη ομάδα επιμηχανική πολιτική με παρουσία του Επιτρόπου Ταγιάννη. Σήμερα έχουμε πάλι την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που συζητά για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν η τυποποίηση και οι σχέσει τη με την επιμηχανική πολιτική είναι πλέον ξεκάθαρη. Τώρα, κάτι που απευθύνεται και προς τον κύριο Ταγιάννη. Είμαστε βέβαιοι ότι η αρχή περί κρατών, μελών και εθνικών φορέων είναι μια αρχή που λειτουργεί για την ώρα, αλλά στο πεδίο του ευρωπαϊκού φορέα τυποποίησης δεν θα πρέπει να τρομάζετε με τις περίεργες ιδέες που ακούγονται για τέτοιο ευρωπαϊκό όργανο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη πρόσβαση, δυνατότητα πρόσβασης για κάποιες ε, για κάποιους από του ενδιαφερομένους για τις τις οργανώσεις, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τις οργανώσεις καταναλωτών και ούτω Ένα σχόλιο, πρόεδρε, οι άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες είναι επίσης κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε σε όλη αυτήν την συζήτηση. Θα αναφέρουμε λοιπόν όσα συζητήθηκαν εδώ στον Επίτροπο Ταγιάννη και Νομίζω ότι μιλήσατε για εναλλακτική γραμμή παραγωγής σε κάποια από τα σχόλιά σας. Επίσης μιλήσατε για τα πρότυπα περί υπηρεσιών. Αυτό φάνηκε να στηρίζεται ευρέω τη συζήτηση σήμερα. Έγιναν σχόλια και από τον Γενικό Διευθυντή για τη διασύνδεση συγκεκριμένων προϊόντων με συγκεκριμένε υπηρεσίε. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα επανέλθουμε σε αυτό και στι διαβουλεύσει μα και πλέον για την ψηφιακή Ευρώπη. Ήδη είπε κάποιο το λόγο το ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία στον τομέα αυτό. Έχετε δίκιο. Οι κοινοπραξίε και τα φόρα δεν μπορούν να μιλάμε την υπόψη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όμω, δεν νομίζω το πρόβλημα είναι τα νομοθετήματα. Μπορεί να υπάρχει ένα νομικό εργαλείο, όπω είπε ο κύριο Σταγιάννη, και ένα τελικά νομοθέτημα να αφορά διάφορου τομεί. Το θέμα είναι πώ συνδυάζονται λοιπόν τα διάφορα νομοθετήματα μεταξύ του και πόσο ευέλικτα είναι. Η ουσία είναι το θέμα και όχι ο αριθμό των ε, νομικών πράξεων. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τη Κομισιόν και γι' αυτό εν τέλει θα δώσω την ατότητα στον Network να λάβει το λόγο για να κλείσει τη συνεδρίαση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την οργάνωση τη τόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ακρόασης. Έντβαρτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Μάλκολμ. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, να πω ότι κανείς δεν αγνοεί τη σημασία των προτύπων, ιδίως αυτό αφορά του εμπειρογνώμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα πρότυπα για την ε, ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τελευταίου μήνε. Είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και να συναντήσω με πάρα πολλού εμπειρογνώμονε, οι οποίοι μερικοί από αυτού είναι εδώ πέρα και επίσης πολλές ευρωπαϊκές οργανώσεις και φορείς και εκπροσώπους μέλη της, ε, των εθνικών φορέων τυποποίησης, εκπροσώπους κομισιών. Όλοι γνωρίζουν το πόσο μεγάλη σημασία που επέχει η τυποποίηση γιατί είναι ακριβώ το έναρσμα για την ανταγωνιστικότητά μα και μα δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το 20 και 20. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που όλοι οι κύριοι παίκτες θέλουν να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία, καλύτερη επικοινωνία για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλοι οι φορείς οι οποίοι είναι ενεργοί στον τομέα αυτό έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εργασία τους. Υπάρχει ένα πολύ καλά οργανωμένο πλαίσιο και δεν θέλουμε να δώσουμε σε κάποιους από αυτούς τους φορείς μεγαλύτερη επιρροή από ότι σε άλλους μίλησε για συνέργειες ο κύριος Ταγιάννη. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας. Φυσικά τα, οι εθνικοί φορείς τυποποίησης έχουν λειτουργήσει πολύ καλά στον τομέα αυτό. Είναι κατά κάποιο τρόπο οι θερμοκοιτίδες της καινοτομίας. Υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, η Sense, Σενελεκ, η έτσι και άλλοι. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν στην τυποποίηση είναι αναντικατάστατος, ιδίως όταν πρόκειται για τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Φυσικά, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη σύνδεση μεταξύ έρευνας, ανάπτυξης, βιομηχανικών στρατηγικών, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Μπέρντον, Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ένα βέλτιστο πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά παράλληλα θα πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο το στόχο της ε, καινοτομία αλλά και τη καλύτερη ρύθμιση, τη μικρότερη γραφειοκρατία, τη πιο αποτελεσματική λειτουργία των αγορών και όμω και του θέματο του κόστου, το οποίο μπορεί να προκύψει από θεσμικέ και οργανωτικέ ανάγκε. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε το κόστος και σε επίπεδο λειτουργικότητος και το κόστος το οποίο επομίζονται οι επιχειρήσεις. Πιστεύω και χρησιμοποιώ τα λόγια του κυρίου Χάρης ότι χρειαζόμαστε δημοσία υποστήριξη. Πιστεύω ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης θα είναι η βελτίωση αυτού του πλαισίου και η επίτευξη των στόχων του 2020. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους και όλους τους συζητητές που ήταν ιδιαίτερα ενεργοί και όλους τους παριστάμενους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε και τους εμπειρογνώμονες για τη συμμετοχή τους. Έχετε τις πληροφορίες, υπάρχει και υλικό απ' έξω αναμένουμε τη συνεργασία μαζί σας. Ακούσα το χρονοδιάγραμμα, δεν θα τα ξαναπώ. Αναμένουμε το πρώτο σχέδιο της έκθεσης Κόζης, Νίκ και βεβαίως θα ακολουθήσει και συζήτηση και όπως βλέπουμε και έτσι θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και φέτος και του χρόνου, οπότε μάλλον θα ξανασυναντηθούμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Λύεται η συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής Βεβαίω θα επανέλθουν στις 4.30 η ώρα γιατί 3 η ώρα υπάρχει η Ολομέλεια για ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 4.30 ώρα θα είναι εδώ ο Υπουργό, ο Ισπανός και η κυρία Γκέπχαρτ για την οδηγία για τις υπηρεσίες στην αίθουσα 1α002 στο κτίριο PHS. Γεια σας, ευχαριστώ.